Αρχίζουμε σιγά σιγά. Καλωσορίζουμε τους ομιλητές και θυμίζουμε στους συναδέλφους ότι η Γιούλεξ στο Κωσυφοπέδιο είναι η μεγαλύτερη πολιτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, λειτουργεί στο Κωσυφο ε, τελευταία τετραετία. Έχει στόχο να ε, βοηθάει και να υποστηρίζει τις ε, αρχές του Κωσυφοπέδιου στα θέματα κράτους δικαίου. Ιδιαίτερα σε θέματα ε, αστυνομίας, δικαιοσύνης και τελωνίων. Η εσωτερική στρατηγική ενθεώρηση που παρουσίασε ο Διευθυντής της ΥΠΣΙΣΗ έχει στόχο να παρουσιάσει τις εξελίξεις ε, και τα γεγονότα στο κοσμοπέδιο και εν ώψη της αναθεώρησης και ανανέωσης της εντολής που λήγει στις 14 Ιουνίου του 2012. Υπάρχουν και επενετικά σχόλια και επικριτικά. Τα μέλη μας θεώρησαν ε, κατάλληλο λοιπόν να διοργανωθεί μια ακρόαση για να εξετάσουμε αυτά τα θέματα. Θα δώσουμε το λόγο στο Διευθυντή Τζεντιλίνη για να μας μιλήσει για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κόσοβο στα πλαίσια της στρατηγικής αναθεώρησης των προσφάτων εξελίξεων στην περιοχή και ε, για τις σχέσεις μας με το Κωσυφοπέδι, ιδιαίτερα το διαρθρωμένο διάλογο για το κράτος δικαίου. Επίσης, ο Διευθυντής ε, Χάμπερ θα μας ε, παρουσιάσει τα βασικά ε, στοιχεία της στρατηγικής αναθεώρησης. Αρχίζουμε με τον Διευθυντή κύριο Τζεντιλίνη. Very Ευχαριστώ πολύ. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Δύο-τρεις παρατηρήσεις έχω να κάνω. Το πιο σημαντικό όμως είναι να θέσουμε αυτή τη συζήτηση στο σωστό πλαίσιο. Και αυτό θα ήθελα να προσπαθήσω να κάνω διότι η EULEX και η αναθεώρησή τη είναι ουσιαστικά τμήμα της ε, συνολικής δέσμευσης που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το κοσυφοπαίδιο. Γι' αυτό θεωρώ ότι καλό είναι να έχουμε μια σαφή εικόνα. Η πρώτη μου παρατήρηση αφορά την ποιότητα των σχέσεών μας με το κοσυφοπαίδιο η οποία θεωρώ ότι έχει βελτιωθεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Απέχει παρασάγκας από αυτό που είχαμε πριν από κάποιους μήνες ή πριν από ένα χρόνο και νομίζω ότι μπορούμε πλέον συλλογικά να προχωρήσουμε στην εφαρμογή της ε, ατζέντα της Θεσσαλονίκης. Ε, και αν δείτε και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, αυτά είναι τα πιο σημαντικά συμπεράσματα στην ιστορία των σχέσεών μας με το Κωσυφοπαίδιο. Περνάμε από την απολευθέρωση των θεωρήσεων διαβατηρίων στις μελέτες ε, σκοπιμών ε, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, πολλή δουλειά μας περιμένει με το κοσφοπέδιο και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το έχουμε κατά νου όταν συζητάμε την Ιούλεξ διότι η Ιούλεξ είναι αναπόσπαστο τμήμα αυτής της σχέσης. Δεύτερη παρατήρηση, η παρουσία μας επιτόπου. τόπου. για να δούμε επακριβώς αυτή τη νέα ποιότητα στις σχέσεις μας. Ε, έχει ενισχυθεί η παρουσία μας στην Πρίστινα, ε, υπάρχει ένας νέος επικεφαλής της αποστολής, η παρουσία της αποστολής είναι ισχυρότερη, πιο αποτελεσματική, εκπροσωπεί καλύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια Ευρωπαϊκή Ένωση που πλέον μιλάμε μία φωνή όλο και περισσότερο. αποχωρούν ε, τα Ηνωμένα Έθνη. Ήταν επιτυχημένη η διαδικασία αυτή και γι' αυτό και υποστήριξε και υποστήριξαν και οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, το όλο θέμα. Και εδώ είμαστε τώρα πλέον στη Γιούλεξ που ε, έχει συνεχή παρουσία και θα το ε, συζητήσουν οι συνάδελφοι λίγο αργότερα, αλλά η πρόκληση είναι να προσαρμόσουμε αυτή την αποστολή στις νέες ανάγκες και στη νέα πραγματικότητα. Ένα τρίτο στοιχείο το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ο διάλογος μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας είναι μια πολύ προσεκτική διαδικασία. Όπως ξέρετε, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει πολλά σε αυτό το διάλογο στο παρελθόν και κατά την άποψή μου αυτό καταδεικνύει ότι μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα και μπορούμε να δούμε ότι το κοσμοπέδιο ρήμασε πολύ. Διότι για να μπορέσει κάποιος να διαπραγματευτεί, να συμφωνήσει και να εφαρμόσει συμφωνίες δεν χρειάζεται μόνο δέσμευση, αλλά χρειάζεται και μέθοδος και οργάνωση και στρατηγική Το τελευταίο έτος λοιπόν μας δίδαξε πολλά. Οι σχέσεις μας λοιπόν, η παρουσία μας, ο διάλογος έχουν γίνει πολλά. Ε, δεν ξέρω αν έχουν γίνει όλα ή αν έχουμε επιλύσει όλα τα προβλήματα. Μάλλον όχι. Είναι πολλές οι προκλήσεις που μας περιμένουν. Ένα-δυο πράγματα να σας πω. Καταρχάς, Νομίζω ότι το κοσυφοπαίδιο θα πρέπει να γίνει όλο ένα και πιο αποτελεσματικό. Οι προσδοκίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το κοσυφοπαίδιο θα αυξηθούν σιγά-σιγά και το κοσφοπέδιο θα πρέπει να μας δίνει όλο και περισσότερα αποτελέσματα και όλο και καλύτερα. Νομίζω ότι αυτός ο χάρτης πορείας για τις θεωρήσεις των διαβατηρίων είναι ένα καλό παράδειγμα. Το είδαμε χθε και αυτός ο χάρτης πορείας σημαίνει ότι θα πρέπει να διπλασιαστεί η προσπάθεια τους προκειμένου να προχωρήσουν. Μια ακόμα πρόκληση, όπως σας είπα, είναι ο διάλογος. Το κοσφοπέδιο και η Σερβία πρέπει να βρουν έναν τρόπο να συνεχίσουν να συνομιλούν για να ομολοποιήσουν τις σχέσεις τους. Ο διάλογος γίνεται για να βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων, να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ Πρίστινας και Βελιγραδίου, για να ε, μην υπάρχουν πλέον προσκόμματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ μακροπρόθεσμο βέβαια αυτό το πρόγραμμα και μπορεί να διαμορφωθεί με διάφορους τρόπους. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση και νομίζω ότι αυτά από πλευράς μου. Σας ευχαριστώ πολύ. The floor has Και τώρα το λόγο έχει ο Διευθυντής κύριος Χάβερ για να μας παρουσιάσει τα βασικά σημεία της στρατηγικής ανθεώρησης. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, την άδειά σας θα είμαι σύντομος. σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της αποστολής και μετά θα σας δώσω μερικές λεπτομέρειες για το γιατί η αποστολή αυτή σε μεγάλο βαθμό χαρακτηρίζεται ως επιτυχής, κάτι το οποίο δεν έχουν γράψει εφημερίδες ως τώρα. Σε ό,τι αφορά την ε, υλοποίηση της στρατηγικής ανθεώρησης για την οποία μιλάμε, ε, υιοθετήθηκε πριν από τρεις μήνες η στρατηγική ανθεώρηση. Ε, το πρώτο σημείο είναι ότι η αποστολή ετοιμάζεται για την μεταφορά ε, εξουσίας ε, και το τέλος της εκτελεστικής εντολής. Μετά από τρία-τέσσερα ε, χρόνια πρέπει να ετοιμαστούμε γι' αυτό. Θα πρέπει να μεταφέρουμε τις αρμοδιότητες μας στις αρχές του κοσμοπεδίου με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και με βάση την πρόοδο που έχει γίνει. Αυτή η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει με όλα τα 20, ε, και, τα 27 κράτη-μέλη έχουν συμφωνήσει. η, η αποστολή αυτή είναι αποστολικά του δικαίου αλλά εστιάζεται, θα εστιαστεί από εδώ και πέρα ε, ακόμα πιο πολύ από ό,τι στο παρελθόν στη δικαιοσύνη. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Τα τελωνία και η αστυνομία έχουν προοδεύσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια στο κοσυφοπαίδιο, όμως ο δικαστικός τομέας ε, ακόμα έχει μείνει πίσω. Θα εστιαστούμε λοιπόν τα επόμενα δύο χρόνια στο, στη δικαιοσύνη, οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά, προστασία μαρτύρων, αλλά και ευαίσθητα διεθνωτικά θέματα όπως περιουσίες ε, και αγνοούμενοι. Υπάρχει βέβαια και το βόρειο Κωσυφοπαίδιο. Η αποστολή έχει μία εντολή για όλη την επικράτεια του Κωσυφοπαιδίου, παρόλο που είναι πολύ πιο δύσκολη η υλοποίησή τη στο βορρά. Οι συγκρούσει για τι οποίε ενημερωθήκατε πέρσι το καλοκαίρι ε, ε οφείλονται στο ότι η αποστολή προσπαθεί να εφαρμόσει τα αποτέλεσμα του διαλόγου, κάτι που εξακολουθεί να είναι μια πρόκληση, ένα πρόβλημα, παρόλο ότι ο διάλογος ε, αυναμένει την επανεκκίνησή του. Ε, πρέπει όμως το κράτος δικαίου να, να αφορά και τον πληθυσμό του Βόρειου σφοπεδίου. Έχουμε μια εσωτερική αναδιάρθρωση της αποστολής από τους τρεις πυλώνες που είχαμε, αστυνομία, τελωνία, δικαιοσύνη, σε μια πιο ε, επιχειρησιακή προσέγγιση πλέον, με δύο πυλώνες. Πρώτον, ενίσχυση δηλαδή ο προηγούμενος μηχανισμός ε, ε, παρακολούθησης και συμβουλών ε, και το, τον εκτελεστικό πυλώνα. Δηλαδή το εκτελεστικό στοιχείο πλέον αποχωρίζεται κατά κάποιο τρόπο. Είναι η τελευταία από τις λειτουργίες που θα αποδοθεί στις αρχές του κοσυφοπεδίου. Όλα αυτά συνοδεύονται από σημαντική μείωση του προσωπικού μας, 25, κατά 25% περίπου, όλοι εσείς που εργάζεστε σε διεθνούς οργανισμούς γνωρίζετε τι σημαίνει μια τέτοια μείωση, τι πρόσθετη προσπάθεια θα απαιτήσει και ότι χρειάζεται και μια μεταβατική περίοδος. Αυτή η μείωση θα μας ε, δώσει αρκετό προσωπικό ελεύθερο για να το ε, ε, χρησιμοποιήσουμε στις νέες μας αποστολές στο Νότιο, στο Νότιο Σουδάν, στη Βόρεια Αφρική κλπ. Όλα αυτά σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της ε, στρατηγικής ε, αναθεώρησης. Τώρα, να σας πω για τις επιτυχίες της αποστολής. Ε, ήμασταν στα πρωτοσέλιδα την περασμένη το περασμένο καλοκαίρι με τις συγκρούσεις στο βόρειο Κωσυφοπαίδιο ε, έγιναν σχόλια και από τον ΝΑΤΟ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποστολή. Αργότερα ε, κάπως σταθεροποιήθηκε η κατάσταση ε, και με και η, μπήκε η Σερβία στο κέντρο της προσοχής, Σερβία και Ευρωπαϊκή Ένωση, εκλογές Σερβία, τέλειωσαν οι εκλογές, καιρός να επανέλθουμε στο Κωσυφοπαίδιο. Θα είναι δύσκολο η αποστολή δημιουργεί προβλήματα σχεδόν σε καθημερινό επίπεδο. Εντάξει, αυτό οφείλεται και στο περιβάλλον βέβαια. Αν μην ξεχνάμε όμως και τις επιτυχίες της αποστολής αυτής. Καταρχήν, ε, βελτίωσε ε, την κατάσταση του Κωσυφοπέδιου. Μετά από τέσσερα ε, χρόνια παρακολούθησης, τα τελωνία στο Κωσυφοπέδιου είναι εξαιρετικά, η αστυνομία γίνεται όλο και πιο επαγγελματική και αναγνωρίζεται αυτό και από τον πληθυσμό όλο και περισσότερο. Συγκεκριμένο παράδειγμα, ε, η παρακολούθηση στο αεροδρόμιο της Πριστίνα ε, μας οδήγησε σε αύξηση κατά 500% σε 12 μήνες ε, σε ό,τι αφορά τα ποσά τα οποία παρανόμως εισερχόντουσαν στο κοσυφοπέδιο. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά το δικαστικό Έχουμε 330 ανοιχτέ έρευνες και περίπου 300 ε, καταδίκες σε ποινικά δικήματα. 330 όπως σας είπα ανοιχτέ έρευνες και περίπου 300 καταδίκες ήδη. 300 δικαστικές αποφάσεις να το πω ε, ε, καλύτερα. Περίπου 200 για ποινικά δικήματα. Ε, ε, έχουμε, το δικαστικό στην έχει αναλάβει πάνω από 1.800, 1800 ε, υποθέσεις. Ε, έχουν διαρευνηθεί πολιτικοί, υπουργοί, ε, ε, επιχειρηματίες, ε, πρώην μαχητές του KLA κλπ. Έχει γίνει επίσης σημαντική πρόοδος στην καταπολέμηση της, ε, της διακίνησης ανθρώπων και οργάνων. Ε, μια σημαντική επιτυχία ε, ήταν η καταδίκη 7 ατόμων για 66 ε, χρόνια με πρόστιμο περίπου 500.000 ε, δολαρίων. ήταν ένα κύκλωμα ε, το οποίο διακινούσε ε, ε, ανθρώπους μεταξύ Σερβίας και Σουφοπεδίου. Επίσης είχαμε και το θέμα των οργάνων. Πέντε άτομα έχουν, δικάζονται αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά το λαθρεμό ναρκωτικών, εισαγγελείς και δικαστές έχουν ολοκληρώσει έξι δίκες σε σχέση με διεθνή δίκτυα. Ε, ποινές μέχρι 15 έτη ε, έχουν δοθεί στους καταδικαστέντες ε, και άλλες 31 περιπτώσεις ερευνώνται αυτή τη στιγμή. Λαθρεμπόριο από κοινού η Γιόλεξ με τα τελωνία του Κωσυφοπεδίου ε, που είναι σε πολύ καλή κατάσταση ε, ε, οδήγησαν σε μείωση του λαθρεμπορίου με εξοικονόμηση εκατομμυρίων ευρώ για το Δημόσιο Ταμείο. Σε ό,τι αφορά την διαφθορά έχουμε έρευνες στο σχέση με το Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών, Μεταφορών και επίση σε θέματα δημοσίων προμηθειών στην αστυνομία ενώ έχει καταδικαστεί ο επικεφαλής του, ε, των, της, ε, των ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνών του Κωσυφοπεδίου. Είχε κατηγορηθεί ε, για απάτη και κατάχρηση ε, θέσης. Τον Μάιο του περασμένου έτους καταδικάστηκαν 8 άτομα για διαφθορά με ποινές φυλάξεις μέχρι 5 έτη. Η υπόθεση αυτή αφορούσε παρατυπίες που εντοπίστηκαν το 2006 στην Credit Bank της Πριστίνα, η οποία έκλεισε κιόλας. Όλα αυτά είναι καλά παραδείγματα για το πόσο μπορεί να κρατήσει μια, η εκδίκαση μιας υπόθεσης, ε, όμως ε, το οικονομικό έγκλημα ε, και, το, και, τα έγκληματα, και, τα έγκληματα πολέμου έτσι κι αλλιώς παίρνουν πολύ χρόνο για να εντοπιστούν ε, και να διερευνηθούν παντού, όχι μόνο στο Κωσυφοπέδιο. Το βλέπουμε και στη Χάγη. Η αποστολή επίση ερευνά εγκλήματα πολέμου. Τον Ιούλιο του 2012 η, ε, ε, ο Σάβιτ Κέτσι καταδικάστηκε και ε, άλλοι τρει για εγκλήματα πολέμου κατά, του, ε, κατά των αμάχων. σε μια άλλη περίπτωση, δύο άτομα καταδικάστηκαν τον Νοέμβριο. Ένας από αυτούς σε 18 έτη φυλάξης για εγκλήματα πολέμου αντίον των αμάχων το 99 και ένας άλλος σε ποινή έξι μηνών με αναστολή για παρόμοια δικήματα. Άλλες, μια άλλη περίπτωση με δέκα ε, κατηγορούμενους είναι η περίπτωση Κλέτσκα, υπόθεση Κλέτσκα. Ένας από αυτούς είναι μέλος του Κοινοβουλίου, πρώην υπουργό. Ε, κατηγορούνται με ε, ανθρωποκτονία ε, και ε, επιθέσεις ε, σε αμάχους και σε ε, κρατούμενους. Για τους αγνοούμενους. Οι ειδικοί της αποστολής έκαναν περίπου 3.000 επιχειρήσεις για για και εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν στις οικογένειές τους τα υπολείμματα 3.000 ατόμων σε ό,τι αφορά το περιουσιακό. αποφασίσαμε επί 23, πάνω από 23.000 ε, ε, αιτήματα επιστροφής περιουσιακών στοιχείων. Ε, ανοίξαμε το δικαστήριο της Δημητρόβιτσα και δημιουργήσαμε και την αιστεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά από όταν άνοιξε το Δεκέμβριο 2008 το δικαστήριο, μετά από 9 μήνες που, ε, χωρίς να λειτουργεί, οι ε, διεθνείς, ε, δικηγόροι, διεθνείς ε, δικαστές και οι εισαγγελίες έχουν ολοκληρώσει 15 δίκες ήδη. Διάλογος Πριστίνα Βελιγραδίου. Όπως σας είπα, η αποστολή εφαρμόζει, υλοποιεί αυτό το διάλογο. Έχουν επιτευχθεί πολλά και θα πρέπει να εφαρμοστούν πια. Όλα αυτά είναι μια συνοπτική παρουσίαση των ε, επιτυχών αποτελεσμάτων της ε, αποστολής. Ας μην τα ξεχνάμε, μόνο και μόνο επειδή αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στο βόρειο Κωσυφοπέδι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις εξηγήσεις σας. Θα παρακαλούσα τώρα ε, τον κύριο Μπούντε Μανάκ που είναι επικεφαλής αντιπροσωπείας στο Κωσυφοπέδιο να μας κάνει τη δική του παρουσίαση. Ευχαριστώ. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Ω συνήθω είναι μεγάλη μου χαρά να παρευρίσκομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να έχω την ευκαιρία να απευθυνθώ στην αξιότιμη επιτροπή σας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ε, να εμπλακεί στο κοσυφοπαίδιο σε σημαντικές διαδικασίες που έχουν σχέση με το κράτος δικαίου, όπως ανέφεραν οι προλαλήσαντες. Ε, εχθές και ο κύριος Φίλερ και η κυρία Μάλστρομ, οι ε, επίτροποι, εγγενίασαν τον επίσημο διάλογο και το διάλογο για τις θεωρήσεις διαβατηρίων για την απελευθέρωσή τους. Εντάσσεται λοιπόν το κοσυφοπαίδιο στην πολιτική μας για τα Δυτικά Βαλκάνια και όπως ε, ακούσαμε προηγουμένως, ε, έχουμε μια νέα στρατηγική, ε, μια συνολική προσέγγιση. Η Γιούλεξ υποστήριξε και θα εξακολουθεί να υποστηρίζει το δρόμο του κοσφοπεδίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βασικό μου μήνυμα σήμερα προς εσάς είναι αυτό ακριβώς. Κάνουμε όλοι συντονισμένες προσπάθειες για να βοηθήσουμε στη συνέργεια και τη συνέπεια των κοινών μας ενεργειών. Μεταξύ άλλων, συνεργαζόμαστε στενά με το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πρίστινα ε, και ε, τον ειδικό επεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους ε, ομολόγους του. Έτσι θα είμαστε σε θέση να συζητήσουμε με το Κωσυφοπέδιο όλα τα θέματα κράτους δικαίου και τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν για την ευρωπαϊκή του προοπτική η αποστολή μας προσβλέπει να συνεργαστεί ακόμα περισσότερο με τις αρχές ε, της χώρας για να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα και την ε, διαφθορά. Είναι μια νέα ευκαιρία ε, και ε, έτσι αναδιατυπώνεται και η αποστολή. Αυξάνονται οι αρμοδιότητες όπως αναφέρθηκε, ιδιαίτερα σε τομείς ε, αστυνομικής συνεργασίας και τελωνίων και μειώνεται το κέντρο βάρους το επιχειρησιακό στην Πρίστινα και στο Βόρειο Κοσφοπέδιο, ενώ διατηρούμε τις δυνατότητες δράσης σε όλο το Κοσφοπέδιο. Αυτό έγινε χάρη στην πρόοδο που έχουν επιτελέσει οι θεσμοί του Κοσμοπεδίου και ε, στα επιτεύγματα της αποστολής. Όπως είπε ο Χαντζιόρκ ε, αριθμητικά, αυτό ε, μας οδηγεί στη δυνατότητα μείωση 25% το στελεχιακό μας δυναμικό. Θα συνεχίσει τη εργασία της αποστολή, αλλά μαζί με την εντολή που ανέθεσαν ε, τα κράτη-μέλη ε, για την επόμενη διετία. Φιλοδοξία η αποστολή είναι, είναι πιο ε, προσαρμοσμένη και συμπληρωματική προς το γενικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κοσυφοπαίδιο και συνεργαζόμαστε με τους θεσμούς κράτους δικαίου της χώρας. Θα εξακολουθήσει η αποστολή να υποστηρίζει την εφαρμογή που χρειάζεται ακόμα, εφαρμογή των συμπερασμών ε, τη διευκόλυνση της ε, υπόθεσης του διαλόγου ε, Πρίστινας Βελιγραδίου για θέματα δημοτολογίου ελεύθερης κυκλοφορίας και η λεγόμενη συμφωνία IBM για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Από την επιχειρησιακή εκτελεστική πλευρά αυτό τι σημαίνει. Αυξάνεται ο αριθμός των ποινικών δικών και των ε, ε, ανακρίσεων και σε επίπεδο αστυνομία και εισαγγελία. Συμφωνούμε τη μεθοδολογία και οι δικαστές ε, του Κωσυβοπεδίου συμμετέχουν σε μεικτά δικαστήρια με δικαστές της Γιούλεξ και αυτά τα δικαστήρια θα είναι αργά ή γρήγορα η πλειονότης. πλειονότη. επιτρεψτε μου να σας πω ποια είναι η φιλοσοφία μας. Είναι απλή. Η αποστολή μας άρχισε με τη βοήθεια προς ε, τις αρχές του κοσμοπεδίου να στήσουν ένα δικαστικό σύστημα ε, και να μπορούν ε, να λειτουργούν με τρόπο αντικειμενικό, αμερόληπτο και χωρίς διεθνή επέμβαση. Τώρα θα επικεντρωθούμε σε θέματα που έχουν σχέση με ε, δίκαιη, διαφανή και βιώσιμη διαδικασία προσλήψεων και ε, άσκηση πολιτικής στο κράτος δικαίου. Έχουμε και μια εσωτερική μονάδα οικονομικής, ε, οικονομικών πληροφοριών και η αστυνομία του Κωσόβου που είναι επιφορτισμένη ε, με τη δίωξη του ποινικού εγκλήματος συνεργάζεται με την εισαγγελία. Το οργανωμένο έγκλημα, η διαφθορά πρέπει να καταπολεμηθούν και ε, έχουν και την προθυμία οι αρχές να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες. Ένα ενισχυμένο νομικό πλαίσιο που θα εφαρμόζεται σωστά και θα δαμάζει τις πολιτικές επεμβάσεις και παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη ε, και θα ε, βοηθάει και στην εκπαίδευση και ενημέρωση των στελεχών υπάρχει ένα πλαίσιο καταπολέμησης της διαφθοράς έτσι ώστε ε, να ε, μειωθεί ε, η διαφθορά και η γενικότερη αντίληψη περί διαφθοράς. Υπάρχει ο διάλογος για τη θεώρηση διαβατηρίων με κάποιους όρους και προϋποθέσεις. Καταλαβαίνετε ότι παραμένει προτεραιότητα αυτή η προσπάθεια με συγκεκριμένους στόχους. Επιτρέψτε μας να σας αναφέρω μερικούς. Η επίτευξη πλήρους ελευθερίας ε, κινήσεων για τη Γιούλεξ και σήμερα πόρο έχουμε. Ε, αύξηση των ε, περιπτώσεων εγκλήματος που οδηγούνται σε δίωξη, ανάκριση και δίκη. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα δίκτυα, το οργανωμένο έγκλημα. Αυτή την εβδομάδα αρχίσαμε αυτή την προσπάθεια. Επίσης, το τοπικό δικαστήριο στη Μητρόβιτσα θα πρέπει να στελεχωθούν οι δικαστικές αρχές και ε, στο βόρειο Κωσυφοπαίδιο να γίνει αντιληπτή και, και αποδεκτή η παρουσία της αστυνομίας του Κωσόβου. Καταλαβαίνετε ε, ότι ε, από το αποτέλεσμα θα κριθεί η Γιούλεξ με συγκριτική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων. Είναι μια νέα εντολή για την επόμενη διετία, αλλά ταυτόχρονα θα χρειαστεί και ένας μηχανισμός εσωτερικής αξιολόγησης ε, benchmarking που να συγκρίνει ε, τα επιτεύγματα με την εντολή και να συμπεριλαμβάνει όλους τους στόχους της Γιούλεξ, ιδιαίτερα προτεραιότητες και δραστηριότητες ε, που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν θέματα εσωτερικών δικαιοσύνης ή διεύρυνσης. Σίγουρα έτσι θα αυξηθεί η προγραμματική αποτελεσματικότητα της αποστολής και ταυτόχρονα θα ε, και θα έρθουν οι συζητήσεις και οι ε, συμβουλές που παρέχονται από τα κράτη-μέλη. Είμαι βέβαιος ότι αυτή η προσέγγιση με βάση το αποτέλεσμα θα οδηγήσει στη γενική επιτυχία της αποστολής και θα προσαρμοστεί το κοσμοπέδιο στα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ως προς το κράτος δικαίου. Και θα είναι μια περαιτέρω ενθάρρυνση των αρμοδίων θεσμών να προχωρήσουν, να επιτελέσουν και μεγαλύτερη πρόοδο για να αναλάβουν και περισσότερες ευθύνες. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Η κυρία Μωρίνα, δεν ξέρω αν το είπα σωστό. Αντζελούσε Μωρίνα, παρακαλώ. Well, me... Λοιπόν, καταρχάς να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου και τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα και μοιραστώ μαζί σας τι απόψει μου επί του ζητήματο. Θα ξεκινήσω με ένα ανέκδοτο. Ζήμε στην εποχή της κοινωνικής δικτύωσης του Facebook και του Twitter και όπως πολλοί από εσά εχθές ενημέρωσα το στάτους μου και τους είπα ότι βρίσκομαι στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχω σε μια κρόαση για τη Γιούλεξ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αμέσως ένας φίλος μου σχολίασε και μου είπε γιατί προσεκλήθη ε, για να μιλήσει για τη Γιούλεξ. Ποιο άλλον θα ρωτούσαν αν δεν ήταν Κωσοβάρος λοιπόν. Και η απάντησή του ήταν ότι η Γιούλεξ δεν είναι κάτι για το κοσυφοπαίδιο, είναι για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Ίσως σήμερα να διαπιστάσουμε ακριβώς για ποιο λόγο βρίσκομαι εδώ και ποια είναι η απάντηση στην ερώτηση. Πέρα από τα αστεία όμως, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το χρόνο που μου δίνεται για να σχολιάσω τρία σύντομα σημεία. Like to uh, the reputation, the image. Καταρχάς, θα ήθελα να μιλήσω για την εικόνα και το παράδειγμα της σταθερότητας και την νοοτροπία αυτή της ατιμορρησίας που επικρατεί στο Κοσμοπέδιο. Το δεύτερο είναι το πώς δραστηριοποιούμαστε, πώς ε, ε βρίσκεται το κόσμο αυτή τη στιγμή, τι γίνεται με τη δικαιοδοσία μας, την αλλαγή του συντάγματο και τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Περιτώ να σας πω ότι το τελευταίο σημείο που θα σχολιάσω είναι το βόρειο κοσφοπέδιο για τη φήμη μας. Είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε καλή ε, φήμη στο... μεταξύ των Κωσοβάρων. Ε, Κάποιοι θεωρούν ότι η αποστολή ήταν ε, απόλυτη αποτυχία, αλλά εγώ συμφωνώ με τις απόψεις που ακούσαμε από τον κύριο Ντερμάρνια και από τον κύριο ε, Χάμπερ. Υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις που όντως μπορούν να θεωρηθούν επιτυχία, αλλά υπήρχαν και πολλές συζητήσεις και δημόσια συζήτηση ε, και σίγουρα η άποψη της κοινή γνώμης ε, κάθε άλλο παραθετική είναι. Ε, κυρίως ε, μας ενδιαφέρει το θέμα σταθερότητα πάνω απ' όλα και ορισμένες περιπτώσεις που διαπιστώσαμε είχαν πολιτικά κίνητρα. Δεν υπήρχαν ουσιαστικές αποδείξεις. Να αναφέρω εδώ την περίπτωση του επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας τον κύριο Ασίμρι Τζέπη, ο οποίος κρατήθηκε για μήνες, βρισκόταν υποκράτηση και τελικώς ε, απελευθερώθηκε γιατί δεν υπήρχαν αρκετές αποδείξεις. Υπήρχαν και κάποιες άλλες περιπτώσεις υψηλού επίπεδου ε, που υπήρχαν θέματα ε, κακοδιαχείρισης, ανικανότητας. Υπάρχει περίπτωση του κύριου Ρακές και την όλη υπόθεση που βασίστηκε σε ένα και μόνο μάρτυρα, το πώς συμπεριφέρθηκαν στο μάρτυρα και το γεγονός ότι ο μάρτυρας δεν βρίσκεται πλέον εν ζωή. Δυστυχώς ε, αυτό το θέμα της ατιμορρησίας εξακολουθεί να μας βαραίνει και η άποψη της κοινή γνώμης στο Κόσοβο είναι ότι αυτό το θέμα ε, διονύζεται. Ε, υπήρχαν περιπτώσεις στις οποίες χάνονταν οι αποδείξεις ε, και δεν ξανακούγονταν ποτέ οι, αποδει... Ε, οι υποθέσεις αυτές, ε, χάνονταν και οι φάκελοι τους και αυτό συνεχίζεται και μέχρι σήμερα. Αυτό βασικά δηλαδή που θέλω να σας πω είναι ότι φαίνεται να υπάρχουν κάποιες υποθέσεις που έχουν πολιτικά κίνητρα και κάποιες από αυτές τις υποθέσεις υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν να εξεταστούν. Ο κίνδυνος λοιπόν ε, της ασφάλειας και της σταθερότητας δεν ε, προκύπτει από τους απλούς πολίτες στο κοσφοπέδιο, διότι οι καθημερινοί πολίτες δεν είναι απειλή για το κράτος δικαίου. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν ε, διάφορα επίπεδα απειλή και κυρίω η απειλή είναι η ίδια η πολιτική, αλλά ε, το βασικό πρόβλημα είναι ότι μπορεί να πέσουμε στην παγίδα και να μην αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στο ανώτερο επίπεδο της πολιτικής. Ε, δηλαδή ε, στα θεσμικά όργανα ε, και εγώ έχω εδώ κατά νου και την ε, δημόσια συμβάσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ στις ε, πέντε χώρες ε, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν μας αναγνωρίζουν. Η διπλωματία της Σερβίας εδώ και χρόνια, από το 2008 και μετά, ε, προσπαθεί από την πίσω πόρτα της Ευρω... των Ηνωμένων Εθνών να μην αναγνωρίσει τη χώρα και αμφισβητεί και τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιείται η αποστολή. Θέλουμε να δούμε τι δυνατότητε έχει η Ευρώπη μετά τη συνθήκη τη Λισαβόνα και πώ μπορεί να καθιδρύσει ένα κράτο δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να στείλει την ε, βασική της αποστολή ε, του κράτους δικαίου σε μια περιοχή στην οποία δεν υπάρχει καθόλου πολιτική για το θέμα. Το, η έννοια της ουδετερότητας της χώρας δυστυχώς είναι λανθασμένη και γι' αυτό το λόγο δεν είναι η σωστή για το κοσυφοπαίδιο. Είτε αναγνωρίζεται είτε δεν αναγνωρίζεται ένα κράτος. Δεν υπάρχει ένα διάμεσο καθεστώς και ε, δυστυχώς αυτό αποτελεί πρόσκομα και δημιουργεί πρόβλημα και δεν υπάρχει κράτος δικαίου σε πολλές περιοχές του Κωσυφοπεδίου. Εδώ θα ήθελα να σταθώ ιδίως στο βόρειο Κωσυφοπέδιο και στην... Ε, ανοχή το γεγονός ότι επιτρέπουμε παράλληλες ε, σερβικές δομές και όχι μόνο στην περιοχή της Μητροβίτσα αλλά και σε άλλες ε, περιοχές. Δεν έχουμε μόνο στο Βόρειο Κοσφοπέδιο. Και υπάρχουν και κάποιες συζητήσεις που λένε ότι θα πρέπει να υπάρχουν ε, αυτές οι δομές διότι παρέχουν υπηρεσίες, κυρίως παιδεία και υγεία. Και αυτό το ακούμε και από ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση καλή είδηση. Ένα δεύτερο στοιχείο για την ουδετερότητα της χώρας και το γεγονός ότι υπάρχουν πέντε χώρες που δεν μας αναγνωρίζουν είναι το θέμα της ε, δικαιοδοσίας και της αλλαγής του συντάγματος που θα πρέπει να γίνει. Ε, περνάμε στην εποχή ε, μετά το ICO την, ε, ε, και θα πρέπει να δούμε την το Διεθνές Πολιτικό Γραφείο και πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Δεν θα πρέπει να αμφισβητηθεί το νέο σύνταγμα στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Εάν κάποιο βρεθεί ενώπιον των δικαστών τη Γιούλε, μπορεί κάποιο να το αμφισβητήσει στο συνταγματικό δικαστήριο του Κωσυφοπεδίου, εάν ε, δεν διευκρινιστεί η βάση ποια νομολογία ε, δουλεύει το Γιούλεξ και μπορεί να υπάρχει και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την ίδια την αποστολή και τις εκτελεστικές αρμοδιότητες. Σήμερα έμαθα ότι αυτές οι εκτελεστικές αρμοδιότητες θα αρχίσουν σιγά σιγά να χάνονται και θα περάσουν σε τοπικό επίπεδο. Αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμία ε, αγωγή για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μία τελευταία μου παρατήρηση για το Βόρειο Κοσμοπέδιο φυσικά. Ξέρετε ότι το κοσφοπέδιο είναι 11.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το 75% είναι γνωστό ως παράδεισος οργανωμένου εγκρήματος ε, διαφθοράς και όλες τις μορφής λαθρεμπόριο. Σε εκείνη την περιοχή ζουν το πολύ 50.000 άτομα. Μετά από το 1999 κανένας δεν κατάφερε να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου σε αυτά τα 1200 ε, τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι μια ελάχιστη περιοχή στην πραγματικότητα. Ε, αν δεν λάβουμε υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα μόνο πέρσι σε 1,7 εκατομμύρια σε θέματα ασφαλείας για τη Λιτινική Αμερική, καταλαβαίνετε πώς είναι η σύγκριση. Μπορεί κάποιο να μου εξηγήσει πώς δεν μπορεί κάποιο να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου σε 1200 τετραγωνικά χιλιόμετρα ή ακόμα και και λιγότερα σε μια μικρή περιοχή του Κωσυφοπεδίου. Πραγματικά θα σα ήμουν ευγνώμων διότι ακόμα και σήμερα δεν καταλαβαίνω πώ γίνεται. Αυτό που χρειάζεται το Κωσυφοπεδίο είναι να το βοηθήσουμε να αποκαταστήσει το κράτο δικαίου στο Βόρειο Κόσοβο. Άκουσα τώρα τον κύριο Ντεμάρνιακ ο οποίο μα είπε ότι η αποστολή του ελπίζει ότι θα τα καταφέρει στο Βόρειο Κόσοβο. Είναι λυπηρό να χρειάζεται η άδεια ε, των ε, κατοίκων ε, για να εξετελέσει κάποιος την αποστολή του. Ολοκληρώνω. Εγώ ως Κωσοβάρα πολίτης αντιλαμβάνομαι ότι χρειαζόμαστε βοήθεια και πρέπει να μας βοηθήσετε αλλά ε, δεν θα πρέπει να μας στέλνετε μία αποστολή σε μία περιοχή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει η ίδια συμφωνήσει για την πολιτική. Εγώ πιστεύω ότι το κοσμοπέδιο μπορεί να δημιουργήσει τους θεσμούς του μόνος του με την κατάλληλη υποστήριξη. Το έχουν καταφέρει κι άλλοι. Ε, οι χώρες της περιοχής τα καταφέρνουν μόνες τους. Και κάποιες και από τις χώρες σας τα έχουν καταφέρει στο παρελθόν. Χρειάστηκε να ξεκινήσουν όλοι εκ του μηδενών. Ίσως μπορούμε και εμείς να τα καταφέρουμε με ελάχιστη υποστήριξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Μωρίνα. Και θα ζητήσουμε τώρα ε, από τον κύριο Χού να μας παρουσιάσει από τη δική σου πλευρά της απόψη. Θα είμαι σύντομος. Γιατί ο υπεύθυνο ότι ε, ε, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση εφαρμογής της στρατηγικής αναθεώρησης Συμφωνώ με τα όσα είπε η προηγούμενη ομιλήτρια. Οι αρχές του κοσυφοπεδίου θα πρέπει να γίνουν, να φτάσουν σε σημείο ώστε να μπορούν να λάβουν οι ίδιες την αρμοδιότητα, τις αρμοδιότητες που έχει η αποστολή. Και αυτό είναι και η, αποστολή ε, της Γιούλεξ. Η διαδικασία ε, είχε σχεδιαστεί πολύ προσεκτικά, λαμβάνοντα υπόψη όλους, τη γνώμη όλων των ενδιαφερομένων, όλων των μερών. Ε, και ήμασταν μπροστά σε σημαντικές εξέλιξεις στο Κωσυφοπέδιο. Για παράδειγμα, αυτά του Ιουλίου, τα γεγονότα του Ιουλίου του 2011, ε, η υποψηφιότητα τη Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόοδο στο διάλογο Πρίστινα-Βελιγράδη και βέβαια εκλογέ στη Σερβία το Μάιο φέτο. Έπρεπε επίσης να λάβουμε υπόψη και την ε, ελευθερία ε, κίνησης. Η αναθεώρηση θα πρέπει να ειδωθεί από αυτό το φως. Η κατάσταση του κοσμοπέδιου είναι δυναμική, αλλάζει μέρα με τη μέρα και μετά από τέσσερα χρόνια παρουσίας θα ήθελα να πω ότι ήδη η αποστολή θα έχει προσαρμοστεί πολύ. Έχει γίνει Πρόοδο και την ανέφεραν οι προομοιολητές. Ε, στα τελωνία οι προδιαφέ έχουν βελτιωθεί δραματικά, δραστικά. Σε ό,τι διαφορά την αστυνομία γίνεται όλο και πιο επαγγελματική. Δεν χρειάζεται να έχουμε προσωπικό σε κάθε γωνία, σε κάθε γοριό, σε κάθε επίπεδο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ακόμα προβλήματα, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχεί την προσπάθειά τη, αλλά χρειάζεται να έχει και μια σταθερή κατάσταση επιτόπου για να βελτιώσουμε, να μεγιστοποιήσουμε τις πιθανότητε επιτυχίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την πιο στενή δυνατή συνεργασία με τις αρχές του Κωσυφοπεδίου. Το Κωσυφοπεδίο είναι ένα κοινό project ε, και θα πρέπει να συνεργαστούμε. Είμαστε σε συνεχή επαφή επίσης με το προσωπικό του ΝΑΤΟ στην, κατά τη διάρκεια ε, της ε, σύνταξης της ε, αναθεώρησης. Ε, έχουμε ενισχυμένη παρουσία στο Κωσυφοπέδιο, ο διάλογος με το ε, Βελιγράδι, ο διαρθρωμένος διάλογος, οι θεωρήσεις, οι συμφωνίες, οι μορικές συμφωνίες, όλες αυτές οι παράλληλες διαδικασίες έχουν προωθήσει ποιοτικά την κατάσταση του κοσυφοπαίδιο και η Γιούλεξ θα πρέπει να προσαρμοστεί και θα το κάνει για να υποστηρίξει περισσότερο αυτό το project. Η στρατηγική αναθεώρηση είχε ως στόχο να αντικατοπτρίσει αυτές τις εξελίξεις και το έκανε. Οι συστάσεις ε, υιοθετήθηκαν από την ε, Πολιτική Επιτροπή ε, φέτος και θα πρέπει να περάσουμε στην εφαρμογή τους. Έχουμε ήδη ξεκινήσει, τα προγράμματα, τα προγράμματα συμφωνήθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Να τελειώσω λέγοντας ότι πρέπει τώρα να ε, εφαρμόσουμε αυτές τις συστάσεις και οι αρχές του κωσυφοπεδίου ε, θα πρέπει να επωφεληθούν της ε, τεχνογνωσίας που έχουν οι δικοί μας και να βοηθηθούν έτσι ώστε κάποια στιγμή να αναλάβουν μόνοι τους στα χέρια τους ε, την ευθύνη αυτών των δράσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Αρχίζει η συζήτηση. Καταρχάς θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Λόνα, Τσέκ, η συγγήτριά μας. Uh, uh, Που μπορεί και να συνοψίσει ακόμα ε, ε, ήδη από τώρα τη συζήτηση. <laughs> Ε, όχι, προφανώς δεν θα συνοψίσω τη συζήτηση. Ε, ερωτήσεις θέλω να κάνω στους προσκεκλημένους. Θα ήθελα να θυμίσω πάλι, ε, ειδικά σε εκείνους που έφτασαν ε, μετά την αρχή της συνεδρίασης, πίσω ε, στο βάθος της αιθούσης θα βρείτε μια φωτογραφική έκθεση με φωτογραφίες που έβγαλε η Γιούλεξ τις περασμένες εβδομάδες ε, έγινε ένας φωτογραφικός διαγωνισμός όπου ζητήθηκε από τους πολίτες του Κουσποπεδίου να στείλουν φωτογραφίες ε, με τίτλο «Εστιάζουμε στον νόμο ε, τα σωστά και τα λάθη». Σας καλώ όλους να δείτε την έκθεση, τις φωτογραφίες, υπάρχει και σχετικό φυλάδιο. Νομίζω ήταν πολύ καλή η πρωτοβουλία αυτή που κάλεσε η Γιούλεξ τους πολίτες της χώρας να δώσουν τις απόψεις τους για το πώς θα πρέπει να είναι η δικαιοσύνη και ο νόμος. Ε, αφού σας είπα λοιπόν αυτό, θέλω να σας ευχαριστήσω για τις δηλώσεις σας. Εγώ είμαι συγγήτρια για το Κόσυφο Πέδιο και παρακολουθώ πολύ στενά τις εξελίξεις, τουλάχιστον την τελευταία τριετία. Πρέπει να πω και εδώ ότι στην αρχή η Γιούλεξ το Κόσυφο ήταν πάρα πολύ ευπρόσδεκτη και δημοφιλής δεν τη θεωρούσαν διάδοχο της Μικ την οποία στο τέλος δεν συμπαθούσαν, ε, θεωρούσαν ότι η Γιούλεξ θα είναι ένα νέο πρόσωπο που θα έρθει να εφαρμόσει το κράτος δικαίου, θα αντιμετωπίσει τη διαφθορά, θα ε, τους ε, ε, φέρει στη δικαιοσύνη και το οργανωμένο έγκλημα. Και όπως η κυρία Μωρίνα έχει ξεθοριάσει αυτή η εικόνα τα τελευταία χρόνια. Και θέλω να ρωτήσω τους προσκεκλημένους μας και τον κύριο Χάμπερ και τον κύριο Ντεμανιά και τον κύριο Χουν. Έγινε στρατηγική αναθεώρηση και είπατε μειώσατε τους αστυνομικούς και τους τελωνιακούς, ε, θα επικεντρωθείτε στη δικαιοσύνη. Ωραία. Σε δύο χρόνια από σήμερα πώς θέλετε να είναι η Γιούλεξ και πώς θέλετε να είναι ε, το δικαστικό σύστημα και η δικαιοσύνη στο κοσυφοπαίδιο. Γιατί όταν μιλάμε για στρατηγική θεώρηση θα πρέπει να έχουμε υπόψη και τους στόχους άλλη ερώτηση. Ανέφερε και κάποιος προηγουμένω. Το θέμα του συντάγματο του κοσφοπεδίου και το θέμα ε, το πότε θα λήξει η ε, ανεξαρτησία ε, υπό επίβλεψη. Κάπως θα πρέπει να εδρεωθεί και ένα πλαίσιο νομικό, συνταγματικό για τους λόγους που ανέφερε η κυρία Μωρίνα. Ένα άλλο ζήτημα το θέμα της ισότητας των φύλων. Στη Γιούλεξ υπάρχει σύμβουλος για θέματα φύλου, πολύ καλό αυτό, ε, να είναι και έτσι στελεχωμένες οι αποστολές αυτές, αλλά μπορείτε να μας ε, ενημερώσετε για το τι έχει επιτευχθεί εκεί. Thing, but also Και στην ίδια τη Γιούλεξ και στη στελέχωση αλλά και στις πολιτικές. Και ένα άλλο ζήτημα που θα με ενδιαφέρει Αναφερθήκατε στη διακίνηση γυναικών στο τράφικινγκ. Έχει εκπαιδευτεί η αστυνομία σχετικά. Οι αστυνομικές μονάδες τώρα της ε, Ulex ε, μειώνονται σε μεγάλο βαθμό. Πώς βλέπετε εσείς αυτό το θέμα της συνεργασίας με την αστυνομία του Παιδίου για ε, το τράφικινγκ έχετε αρκετό προσωπικό για να εκπαιδεύετε και τους ε, αστυνομικού του κοσυφοπεδίου ή μήπως θα επέλθουν προβλήματα από τη μείωση ε, των ε, στελεχών σας. Άλλο θέμα. Επανειλημμένα αναφερθήκατε στον κύριο Λίμαη που ήταν μία από τις πολύ γνωστές περιπτώσεις στο κοσυφοπέδιο και με μεγάλες προσδοκίες να καταδικαστεί. Σήμερα ούτε η ε, υπόθεση για το έγκλημα πολέμου, ούτε η υπόθεση για το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά έχουν προχωρήσει. Και αυτό έχει απογοητεύσει πολλού στο Κωσυφοπαίδιο και το έχω ακούσει από πολλού. Βέβαια, εμεί δεν ε, είμαστε εδώ για να παρεμβαίνουμε στη δικαιοσύνη, αλλά πώ εξετάζετε και αντιμετωπίζετε εσείς αυτές τις υποθέσεις. Ξέρουμε ότι πολλές υποθέσεις έχουν ε, τέλες ειδικής με καταδίκες, αλλά ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται έτσι στο κοσυφοπαίδιο. Είναι μεγάλες οι προσδοκίες και οι ελπίδες που δημιουργήθηκαν, ε, αλλά οι ρυθμοί που ακολουθούνται δεν είναι ε, αρκετά ταχύ. Και ξέρω από τη χώρα μου την Αυστρία ότι οι περιπτώσει διαφθοράς είναι δύσκολες στη διερεύνησή του και χρειάζονται χρόνο. Δεν το αγνοώ, δεν το παραγνωρίζω, αλλά στο κοσυφοπαίδιο αυτέ όλε οι ελπίδε και προσδοκίε θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Αυτή ήταν η ε, ερώτηση και το τελευταίο. Το, η ουδετερότητα ω προς το Καθεστώ. Η Γιούλεξ είναι σημαντική αποστολή και χαίρομαι που συμμετέχουν και την υποστηρίζουν, εν πάση περιπτώσει, και 27 χώρες μέλη. Αλλά σε θέματα περιουσιακά, οι δικαστές και οι εισαγγελείς οι ίδιοι αποφασίζουν ποιο νομικό σύστημα ε, θα εφαρμοστεί. Της πρώην Ιουκοσλαβίας, της Ούνμικ ή νόμος του Κωσυφοπεδίου. Εγώ πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει και με την έλλειψη πολιτικής βούλησης η πολιτική συνοχή στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να πούμε ότι είναι κράτος αναγνωρισμένο το κοσυφοπαίδιο και έχει και ε, σύστημα ε, δικαίου. Ξέρω ότι είναι δύσκολο για σας γιατί υπάρχει ουδετερότητα ως προς το καθεστώς του κοσυφοπαιδίου και δεν το υποστηρίζουν πλήρως όλα τα κράτη-μέλη. Προστασία των μαρτύρων. Νόμος υπάρχει. Δεν εφαρμόζεται, αλλά υπάρχει. Και ένα μέρος του προβλήματος είναι ότι τα κράτη όχι μόνο τη Ένωση, αλλά και άλλα κράτη που συμμετέχουν στη Γιούλεξ, εξ όσων κατανοώ εγώ, δεν είναι πρόθυμα να ε, βοηθήσουν στην επαναγκατάσταση των μαρτύρων, δηλαδή να βγάλουν κάποιου ανθρώπους από τη χώρα και να τους ε, προστατεύσουν στη δική του επικράτη. Τα κράτη-μέλη της Ένωσης συνεργάζονται με τον τρόπο που εσείς θα θέλατε. Επίσης δεν βοηθούν ε, δικαστές και εισαγγελείς ε, τα κράτη-μέλη. Δεν αποσπούν δικούς τους δηλαδή εκεί. Και ένα τελευταίο. Αφού παρευρίσκεται και ο κύριος Δεμανιάκ. Ε, λίγη εντολή σας δυστυχώς. Έχει ληφθεί απόφαση για τον αντικαταστάτη σας για την επικεφαλής εκεί της αποστολής. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Chairman. Also... Και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Ακούμε ότι αλλάζει η εντολή της Γιούλεξ. Θα είμαι λίγο έτσι προκλητικός, αλλά ε, αυτό είναι από αποτέλεσμα της αλλαγής της κατάστασης επιτόπου, αν ναι, τι έχει αλλάξει ή μήπως αυτή η αλλαγή ακολουθεί το συμπέρασμα της αναθεώρησης ότι η γιουλεξ δηλαδή ε, δεν πληρεί, δεν επιτυγχάνει πλήρως τους στόχους της στο κοσυφοπέδιο. Τώρα σε ό,τι αφορά το βόρειο κοσυφοπέδιο. Πώς λειτουργούν τα δικαστήρια στο βόρειο κοσυφοπέδιο και τι μπορεί να βελτιωθεί εκεί. Ποια είναι επίσης η πραγματική κατάσταση στις, στα δύο ε, συνοριακά φυλάκια ε, σε ό,τι αφορά τους αστυνομικούς και τελωνικούς ελέγχους. Πότε περιαναμένουμε ότι αυτοί οι έλεγχοι θα αποδοθούν ξανά στις αρχές του που τελειώσουν. Τώρα, διαφθορά σε υψηλά στάμενα πρόσωπα. Στο παρελθόν Έχω την εντύπωση ότι η Γιούλεξ ήταν πολύ γενναία, αλλά μετά σαν να φοβήθηκε από όσα είχε κάνει και όλα άρχισαν να θαμπώνουν, να θολώνουν. Η κυρία Μωρίνα ήταν ε, πολύ διπλωματικά, είπε ότι η Γιούλεξ δεν είναι πολύ δημοφιλή στο κοσυφοπαίδιο. Όταν ε, μιλάμε με τις ε, μη κυβερνητικές εκεί και ταξιδεύουμε εκεί ε, βλέπουμε ότι οι επικρίσεις είναι πάρα πολύ ισχυρές. Ακούσαμε τις εξηγήσεις του κ. Ντεμαρνιάκ ε, και ελπίζουμε ότι θα αλλάξει η κατάσταση. Θα μπορούσατε επίσης να μας δώσετε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες ε, για τις έρευνες του, με βάση την έκθεση του Dick Martin. Ευχαριστώ την κυρία Μωρινά γιατί ε, μας άνοιξε καινούριου ορίζοντες ως, όπου, ως προς το πώς βλέπουμε το ρόλο της Γιούλεξ εκεί. Ευχαριστούμε κύριε Κούκαν. Ο λόγος του κύριο Πόσελτ. Παρακαλώ πολύ δύο λεπτά στον καθένα. Κύριε Πρόεδρε, δεν συμφωνώ να βάζουμε τέτοιους κανόνες μεσούς στις συζητήσεις. Από την αρχή, αν θέλετε, κανόνες. Ε, θέλω να κάνω μια παρατήρηση στην κυρία Μωρίνα τη συγχαίρω για το θάρρος της. Μπορώ να υπογραμμίσω ε, κάθε πρόταση που είπε και θα πρότεινα στην επόμενη ακρόαση να φέρουμε επικριτές ε, και ε, από την τοπική αυτοδιοίκηση και πολίτες του Κωσυφοπεδίου να μας τα πούν. Έχω τρεις συγκεκριμένε ερωτήσεις. Πρώτον, στον κύριο Χάρμπορ. Χάρπερ, συγγνώμη. Τι λέτε για τις κριτικές που ακούμε από την gay ότι μεγάλοι διεθνείς εγκληματίες εντοπίζονται στο βόρειο κοσυφοπέδιο και μετά δεν μπορεί η Γιούλεξ ε, να πάει να τους συλλάβει σε κάποιο λογικό διάστημα, δηλαδή μέσα σε 8-10 ώρες και μετά αυτοί πάλι ε, διαφεύγουν τη σύλληψη και φεύγουν από εκεί. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπούντε Μαρνιάκ. Εφόσον υπάρχουν παράπονα και καταγγελίες που υπάρχουν πολλά στη χώρα, δεν ξέρω αν είναι θεμητά ή όχι. Πρώτον, ποιες δυνατότητες έχει κανείς στο ιστορικό της Γιούλεξ να καταθέσει καταγγελίες και παράπονα και ποιες εκτός. Δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ε, ε, Γιούλεξ. Και τρίτη και τελευταία ερώτηση στον κύριο Τζεντιλίνη. Θέλω να σας ρωτήσω, μετά την εφαρμογή της συμφωνίας που ε, έχει κάνει την κυρία Ταγέρ με τους ε, Σέρβους. Βέβαια μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί τίποτα. Τι γίνεται ε, για την επιτάχυση και τι γίνεται με την εμπορική συμφωνία με το Κωσφοπέδιο. Δεν ακούσαμε τίποτα. Και ένα τελευταίο. Και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει τώρα να ασκήσουμε πίεση ως Κοινοβούλιο. Ανταποκρίνεται αυτό και στα δικά μας ψηφίσματα. Τα κράτη-μέλη που δεν έχουν αναγνωρίσει το Κόσοβο επιτέλους να το αναγνωρίσουν γιατί έτσι διευκολύνεται το έργο και των δημοκρατικών θεσμών ε, του Κωσόβου ε, αλλά και ε, της Ιούλεξ που σε αντίθετη περίπτωση προφανώς δυσκολεύεται. Ο κύριος Παντζέρη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, θεωρώ δεδομένο ότι χρειάζεται δουλειά για να κάνει βήματα προς το μέλλον το κοσφοπέδιο και να έχουμε μεγαλύτερη περιφερειακή ολοκλήρωση και καλύτερη προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναλάβει τα ενία του μέλλοντό του το ίδιο το Κόσοβο. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ξανασκεφτούμε λίγο καλύτερα αυτή τη στρατηγική αναθεώρηση η οποία καθόλου δεν με πείθει η ανανέωση της αποστολής θα πρέπει να προκύψει μετά από μια πιο εις βάθος ανάλυση. Θα πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός, επιχειρήσεις, διαχείριση, ε, επιθε, εποπτεία του ε, Γιούλεξ, να δούμε και γιατί δεν έχουμε καθόλου ικανοποιητική απόδοση μέχρι τώρα. Όλα αυτά βέβαια για να επιτύχει η μελλοντική αποστολή. Η άποψή μου είναι ότι υπάρχουν και κάποιες διαρθρωτικές ελλείψεις οι οποίες θα μπορούσαν να διορθωθούν αν δούμε καλύτερα την κατανομή των πόρων της Γιούλεξ, τον προπολογισμό της, την επιλογή του προσωπικού, ε, τις αποζημιώσεις τους και τη διάρκεια των συμβάσεών τους και να ενισχύσουμε και το σύστημα εσωτερικής ευθύνης αλλά και το σύστημα εποπτείας από πλευράς Βρυξελών. Νομίζω ότι η Γιούλεξ θα πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει πολιτικό ρόλο και να προσέχει και να είναι και ιδιαίτερα διεξοδική ε, στα όσα γίνονται εσωτερικό στο κοσυφοπαίδιο. Αλλά για να γίνουν αυτά ε, ο ρόλος της δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στον άξονα της δικαιοσύνης, αλλά θα πρέπει η δικαιοσύνη να διαχωριστεί και από το πολιτικό σκέλος για να υπάρχει ανεξαρτησία του δικαστικού τμήματος. Δεν μπορεί δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι που μιλούν για πολιτική και σταθερότητα με τον Πρωθυπουργό του Κωσυφοπεδίου και με τους ειδικού εκπροσώπους και τους πρέσβεις και οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι να αποφασίζουν από εκεί και πέρα για τη συμβόλαια των δικαστών και των εισαγγελέων. Επομένως, καλώς μεν να υπάρξει μια καλύτερη ισορροπία και να περάσουμε από τον έλεγχο των συνόρων και των τελωνίων στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση για την ανεξαρτησία του δικαστικού τμήματος και υπάρχουν και κάποια θέματα στα οποία θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Οι σχέσεις με την πολιτική ελίτ του Κωσυφοπεδίου. Θα πρέπει και εδώ να εξευρεθεί μια ισορροπία μεταξύ της αναγνώρισης κάποιων θετικών στοιχείων και της τιμωρίας της λανθασμένης συμπεριφοράς ε, αυτής της πολιτικής ελέητ με συγκεκριμένες πράξεις. Επίσης θα πρέπει να γίνει και κάτι με το, για το θέμα της διαφθοράς, αλλά θα πρέπει να εξισορροπήσουμε και πάλι ε, τις δραστηριότητές μας, διότι μέχρι τώρα έχουμε επικεντρωθεί στα εγκλήματα πολέμου και λιγότερο στη διαφθορά και στο οικονομικό έγκλημα και θα πρέπει να σταθούμε και σε αυτή τη συνιστόσα. Και τέλος θα πρέπει να σταθούμε περισσότερο στις εκτελεστικές αρμοδιότητες και όχι μόνο ε, στα θέματα ε, τα πιο απλά, τα οποία είναι λιγότερο επικίνδυνα μεν και πολύ πιο εύκολα, αλλά θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται σε εκτελεστικό επίπεδο. Ε, και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κατά πόσον γίνεται με την κατάλληλη ποιότητα η κατανομή των πόρων. Πρέπει όμως να γίνει μια καλύτερη αναθεώρηση, γιατί αυτή η στρατηγική αναθεώρηση δεν αρκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Παντσέρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω σλοβενικά καλύτερα στη συζήτηση αυτή. Ωστόσο, πρέπει να αναγνωρίσω ότι έχω πολύ καιρό να πάω στο Κωσυφοπέδιο και δεν γνωρίζω πολύ καλά την κατάσταση του σύνεγγης. Ε, παρόλο αυτά που ακούσαμε σήμερα, είναι πολύ πιο εύκολο να επικρίνουμε τη Γιούλεξ παρά να την επενέσουμε. Όλα αυτά, θέλω να πω ότι διαδραμάτισε ε, σπουδαίο ρόλο και επιτέλεσε μεγάλο έργο η Γιούλεξ σε μια επικράτεια όπου το κράτος δικαίου δεν έχει πολύ μεγάλη παράδοση. Πολλές φορές είχαμε ε, πολλά και διάφορα αντιφατικά φαινόμενα στην ε, περιοχή. Πήγα πρόσφατα σε μία περιοχή και διαπίστωσα ότι ε, η διεισόμαση ότι το Κωσυφοπαίδειο με τη βοήθειά μας πρέπει να κάνει περισσότερες προσπάθειες για το μέλλον, για τους πολίτες του. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω την εξή ερώτηση. Επενδύουμε σε ανθρώπινο δυναμικό στο κοσυφοπαίδιο, στο συγκεκριμένο τομέα το δικό σας. Το κοσυφοπαίδιο θα είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του ε, και να ε, μπορέσει να διαχειριστεί ο ίδιο, το ίδιο τα θέματα κράτους δικαίου. Δυστυχώς, το μέλλον του κοσφοπεδίου εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό και από τη στάση της Σερβίας. Γι' αυτό και θεωρώ ότι το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σερβία είναι ενθαρρυντικό. Μπορεί να μας οδηγήσει σε μεγαλύτερη ισορροπία ε, στις σχέσεις με το κοσφοπέδιο, αλλά αυτό συνεπάγεται και μεγαλύτερη ευθύνη. Η Σερβία βέβαια θα πρέπει και η ίδια να λάβει μερίδιο της ευθύνης, αλλά αυτό θα γίνει μόνο εάν επιμείνουμε και εμείς ότι η Σερβία έχει κάποια ευθύνη όσον αφορά το ευρωπαϊκό της μέλλον και την ευρωπαϊκή της προεπτική. Και ολοκληρώνοντας κύριε Πρόεδρε, διαφωνώ να μας περιορίζετε το χρόνο ομιλίας. Πέντε συνάδελφοι είμαστε όλοι και όλοι. Θα έπρεπε να έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τάνοκ. Συγγνώμη, κυρία Πακ. Δεν μίλησε ο κύριο Τάνοκ, ο κύριο Βάικελ. Α, τώρα πρώτο ο Τάνοκ, λέει κυρία Πακ. Τα τελευταία 11 χρόνια ε, ε, ε, μάλλον ε, πρόσφατα ε, μου ε, ήρθε στην, στην γραφεία μου κάποιος ο οποίος κατήγγειλε ε, προβλήματα με, ε, με τις, τα ορυχεία ε, που έχουν δύο σκέλη, ένα στο βορρά και ένα στο νότο. Ε, το βόρειο σκέλος της ε, εταιρείας ε, υποφίσταται σημαντικά, σημαντικούς περιορισμούς από την Πριστίνα σε ό,τι αφορά το φορολογικό του καθεστώς ενώ το νότιο κομμάτι δεν αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα. Η Ulex δεν αρνήθηκε να ερευνήσει την περίπτωση ή να επιβάλλει πίεση στην κυβέρνηση του Κωσυφοπεδίου. Αυτό ε, καταδίκασε την εταιρεία αυτή στο βόρειο Κωσυφοπέδιο και έμειναν 3.500 άτομα χωρίς δουλειά. Ε, το νομικό καθεστώς της εταιρείας ε, αυτή τη στιγμή εκκρεμεί μέχρι να ρυθμιστεί το συνολικό καθεστώς του Κωσυφοπέδιου. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Δεν θα ήταν καλύτερο η Γιούλεξ να επαναφέρει το καθεστώς που λειτουργούσε για 11 χρόνια παλιότερα. Μετά, οι εκλογές στη Σερβία και ο νέος πρόεδρος ε, που προέρχεται από εθνικιστική παράταξη. Πιστεύετε ότι θα δυσκολέψει την εργασία, το έργο της Γιούλεξ. ή θα συνεχιστεί μια ρεαλιστική προσέγγιση όπως το παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα κυρία Πάκ, Ευχαριστώ Πρόεδρε για τη δυνατότητα που έχουμε σήμερα ε, να συζητήσουμε με τους ε, κυρίους και τις κυρίες. Θα ήθελα να πω ταξίς για τη Γιόλεξ. Μετά την ατυχή μακροχρόνια περίοδο της UNMIC, οι ελπίδες ε, αποτέθηκαν στη Γιούλεξ και μάλιστα μεγαλύτερες από εκείνες που μπορούσε να υλοποιήσει. Ε, ε, πάντα γίνεται αυτό. Μας άφησε το Κόσοβο η Γιούλεξ σε κακή κατάσταση και ήταν δύσκολο να βελτιωθούν τα πράγματα. Θα μπορούσε η Γιούλεξ να είναι πιο αυστηρή σε ορισμένα πράγματα. Βέβαια, όποιος είναι έξω από το χορό πολλά τραγούδια ξέρει ε, και είναι δεδομένα τα εργαλεία που έχουμε. Εγώ θα επιθυμούσα η Γιούλεξ να μπορεί να συνεργάζεται περισσότερο με την K4 ε, για να επιβληθεί περισσότερο το κράτος δικαίου και να προβληθεί ιδιαίτερα στο Βορρά. Κάτι όμως που με ενοχλεί ιδιαίτερα και με εξοργίζει είναι ότι ο διάλογος μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου που άρχισε πέρσι γιατί οι Σέρβοι θέλουν να πάρουν το καθεστώς υποψήφιας χώρας ε, δεν οδηγήθηκε ε, σε αίσιο πέρας. Υπήρξαν αποτελέσματα γιατί δεν είδα εγώ. Ε, και είναι και πολύ αμφίβολα αυτά. Μήπως η Γιούλεξ θα πρέπει και μπορεί να επέμβει περισσότερο σε αυτό. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Για το Βόρειο Κωσυφοπαίδιο. Κατά την άποψή μου, και όχι μόνο τη δική μου, τα λένε και άλλοι που γνωρίζουν περισσότερα από μένα γιατί πηγαίνουν συχνά εκεί, η μαύρη τρύπα εγκληματιών είναι. Και ρωτώ, αυτό το δίκτυο είναι μόνο Σέρβοι εγκληματίες ή μήπως υπάρχουν και άλλοι εκεί ε, που κανονίζουν πολύ ωραία τις δουλειές τους, Αλβανείς ε, καταγωγής εγκληματίες ε, και κρύβονται πίσω από τους Σέρβους. Δεν μπορείτε πια να καθαρίσετε αυτό το λάκκο με τα φίδια τα εγκληματικά. Εγώ ε, είμαι πρόεδρος μιας επιτροπής που ασχολείται και με άλλα θέματα. Γιατί δεν μπορούν οι αθλητές του Κωσυφοπηδίου να πάνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες με τη σημαία του Κωσόβου. Είναι έσχος και ντροπή απέναντι στους νέους, στη νέα γενιά. Σήμερα δεν έχει ε, παραβιάσει κανένα διεθνές δίκαιο το Κωσυφοπέδιο όταν κήρυξε την ανεξαρτησία του. Την ανακήρυξε. Ε, είναι λίγες οι χώρες που δεν το έχουν αναγνωρίσει. Ελπίζω γρήγορα να το αναγνωρίσουν. Είναι κρίμα, έσχος, ντροπή και όνειδος απέναντι στους νέους. Και θα ήθελα να παρακαλέσω και τη Γιούλεξ και τον κύριο Τζεντιλίνη να κάνετε ό,τι μπορείτε. Να υπάρξει ένα φως στην άκρη του τούνελ. Να μην επικεντρωνόμαστε μόνο στα πολιτικά. Και ένα τελευταίο. Αν υπάρχουν εδώ αμφιβολίες στο Κοινοβούλιο, για το αν μπορούμε να αφήσουμε την ανεξαρτησία στα χέρια του κοσφοπεδίου. Ε, να μην επαναλάβουμε το λάθος που έγινε στη Βορζία Ερζεγοβίνη. Όσο κρατούμε κάποιον εκεί επιτόπου ε, περισσότερο που έχει τον τελευταίο λόγο, τόσο λιγότερο αναλαμβάνει τις ευθύνες του ο τοπικός πληθυσμός. Στο Κόσοβο οι άνθρωποι δεν είναι πιο ανόητοι από όπου αλλού και πολλοί ε, που κατέχουν υψηλά ηγετικά ε, αξιώματα, έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό ή ακόμα και στην Πρίστινα, είναι πολύ μορφωμένοι και αξιόλογοι και να τους εμπιστευόμαστε και να μην πάμε εκεί και να τους κουνάμε το χέρι ως δάσκαλοι, να τους βοηθήσουμε, αλλά να τους βοηθήσουμε να βοηθηθούν οι ίδιοι και να αναλάβουν τις τύχες τους. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πακ για τα σημαντικά αυτά σχόλια. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας για να απαντήσουν στις παρεμβάσεις των μελών της Επιτροπής. Πρώτα ο διευθυντής κύριος Τζεντιλίνη. Παρακαλώ. Um, Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Ένα-δυο σχόλια για τις ερωτήσεις που απευθύνθηκαν σε μένα και εν γέννη για τη συζήτηση. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι ότι νομίζω ότι η συζήτηση αυτή και τα πολύ εύστοχα ερωτήματα που ετέθησαν αποδεικνύουν πόσο περίπλοκο είναι το έργο μας, πόσο περίπλοκα είναι τα καθήκοντα που έχουμε αναλάβει. Όλοι όσοι ασχολούμαστε με το κοσυφοπαίδιο. Σίγουρα και μπορούμε να τα πάμε καλύτερα. Ε, ε. Αλλά για την περίπτωση της Γιούλεξ κατά την άποψή μου, πολύ συχνά υπήρχαν πολύ συγκεκριμένε περιπτώσεις οι οποίες κατά κάποιο τρόπο επεσκίασαν τις πολύ περίπλοκες ε, έντονες και δύσκολες καθημερινές ε, δραστηριότητες ε, της Γιούλεξ στο Κοσμοπέδιο κάθε μέρα και το γεγονός ότι παρήχθη έργο αναγνωρίζεται από το γεγονός ότι υπήρξε αναθεώρηση ε, και αναγνωρίζεται και από το γεγονός ότι όπως έλεγε και η κυρία Πακ προηγουμένως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αναλάβουν ε, οι Κωσοβάροι όλο ένα και περισσότερες ευθύνες και να τα καταφέρουν μόνοι τους και μπορούν να τα καταφέρουν και το έχουμε διαπιστώσει όλοι. Και νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή άγουσα. Τώρα, για το διάλογο το είπα ήδη, ελπίζω να κατανοήσουν όλοι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Σαφώς και υπάρχουν οι συμφωνίες, ε, θα σταθώ σε αυτό εντός ολίγου, αλλά θα πρέπει να επισημάνω πόσο σημαντική είναι και η μέθοδος. Η μέθοδος αυτή, όπως σας είπα, ήταν αυτή που ήταν αποτελεσματική και μπορούμε να μάθουμε πολλά από αυτό. Όπως σας είπα, ε, μπορεί να λάβει διάφορες μορφές ε, το όλο θέμα στο μέλλον, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε μέθοδο. Και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Οι συμφωνίες τώρα γίνονται για να εφαρμόζονται. Αυτό είναι γεγονός και θα πρέπει να το τηρήσουμε. Κανείς ε, νομίζω δεν είναι ικανοποιημένος από το ρυθμό με τον οποίο ε, προχωρά αυτή η διαδικασία εφαρμογής, αλλά ε, συνεχίζουμε να πιέζουμε, διότι όπως σας είπα, οι συμφωνίες γίνονται για να εφαρμόζονται. Κάποιες από αυτές τις συμφωνίες έχουν εφαρμοστεί. Κάποιες από αυτές τις συμφωνίες έχουν οδηγήσει αποτελέσματα. Για παράδειγμα, για τα τελωνιακά ζητήματα νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Ελευθερία ε, α, μετακίνηση αγαθών, ελευθερία ανθρώπων. Υπάρχουν αυτά αποτελέσματα. Ε, υπάρχουν κάποια παραδείγματα. Υπάρχουν βέβαια και τομεί στους οποίους ακόμα πρέπει οι δεσμεύσεις να μεταφραστούν σε πράξεις. Και οι δύο πλευρές ε, ε, πρέπει να μεταφράσουν τις δεσμεύσεις τους σε πράξη. Συμφωνώ όμω και με την κυρία Πακ. Υπάρχει φω στην άκρη του τούνελ και νομίζω ότι ο μόνο δρόμο είναι να συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά. Δεν είναι εύκολο, όλα όσα σχετίζονται με το κοσφοπέδιο είναι περίπλοκα. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι να είμαστε ε, επιποδός, να δείξουμε τη δέσμευσή μας και να προχωρήσουμε. Και κάποια στιγμή θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τζεντιλίλη και τώρα ο κύριος Χάμπερ. Μην ξεχνάμε ότι η Γιούλεξ είναι μια αποστολή κράτους δικαίου. Δεν είναι αποστολή με εξουσίες του κεφαλαίου 7 σε ε, περιβάλλον μετασυγκουσιακό. Στόχος της είναι να βελτιώσει τις προδιαφέρειες του κράτους δικαίου στο κοσυφοπαίδιο με μη στρατιωτικά μέσα και με εκτελεστικές εξουσίες περιορισμένες στο δικαστικό σύστημα. Ένα μέρος της έλλειψης δημοφιλίας της Γιούλεξ στο Κωσυφοπαίδιο και της ε, απογοήτευσης από πλευράς του τοπικού πληθυσμού ε, παρόλες τις επιτυχίες που σας ε, περιέγραψα οφείλεται στο ότι υπήρχαν υπερβολικές προσδοκίες. Μετά από 8 χρόνια της Γιούνμικ Είχε ήδη δημιουργηθεί ε, απογοητεύσει στο Κωσυφοπέδιο για μία επιτυχία των στόχων και περίμεναν θαύματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι διχασμένη σε ό,τι αφορά την αναγνώριση του Κωσυφοπέδιου και αυτό ε, αντικατοπτρίζεται και στην αποστολή. Εμείς θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη. Γιατί η αποστολή είναι αποστολή του Συμβουλίου. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε εμείς αυτό. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να το αλλάξουν. Εμείς καταδεικνύουμε τις συνέπειε αυτής της συμφωνία για τις πρακτικές, για την πρακτική λειτουργία τη αποστολή. Το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αλλάξει την κατάσταση. Σε ό,τι αφορά την ε, δικαιοσύνη και τις διάφορες υποθέσεις. Πράγματι, οι προσδοκίες ήταν πολύ ψηλέ στην αρχή. Δεν είναι δυνατόν να... Οι, οι, εύκολες γρήγορες επιτυχίες δεν είναι εύκολες. Μιλάμε για διαφορά, μιλάμε για ε, εγκλήματα πολέμου. Θυμηθείτε τα εγκλήματα πολέμου μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πόσο καθυστέρησαν να τιμωρηθούν. παρόλα αυτά, σιγά σιγά προχωράμε. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξο. Χωρίς να θέλω να είμαι και παράλογος. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξο γιατί αυτές οι υποθέσεις καθυστερούν δύο-τρία χρόνια στη διερεύνησή τους πριν ξεκινήσει η ακροματική διαδικασία. Οπότε ε, δεν μας εκπλήσει ότι δεν είχαμε σημαντικές επιτυχίες το, τα πρώτα πρώτα χρόνια. Ε, όμως όλο και περισσότερες υποθέσεις οριμάζουν. Ασφαλώς και υπάρχει κακοδικία πολλές φορές για παράδειγμα, στην περίπτωση του κυβερνήτη της Κεντρικής Τράπεζας, του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, ε, υπάρχουν άλλες υποθέσεις στις οποίες οι, ε, οι αμάρτυρες πεθαίνουν, όπως στην περίπτωση του κ. Λιμάη. Ε, ο θάνατος και σαν και άλλες είναι από φυσικά αίτια ή ατύχημα. Αυτό όμως δεν είναι αντεπιχείρημα για αυτούς που προσπαθούν να φέρουν αυτές τις υποθέσεις στο δικαστήριο θα πρέπει να δεχτούμε αυτό το κομμάτι, αυτά τα ατυχήματα, ως τμήμα του δικαστικού συστήματος. Ε, δεν πρόκειται να υπαναχωρήσουμε έναντι των υψηλών στάνταρ που έχουμε θέσει για τη δικαιοσύνη. Δεν μπορώ να σχολιάσω την ουδετερότητα σε ό,τι αφορά το καθεστώς από πλευρά μα. Αυτό είναι μια αρχή η οποία μας έχει επιβληθεί από τα κράτη-μέλη. Ένα άλλο θέμα ήταν η προστασία των μαρτύρων. Χρειαζόμαστε την προστασία των μαρτύρων και χρειαζόμαστε προσωπικό για την προστασία των μαρτύρων. Δεν έχουμε πολύ προσωπικό. Δεν μα έχουν στείλει πολύ προσωπικό τα κράτη-μέλη. Οπότε ε, εξακολουθούμε να το ζητάμε. Και επίσης εξακολουθούμε να ζητούμε την επανεγκατάσταση των μαρτύρων. Και πάλι όμως διστάζουν τα κράτη-μέλη. Ρωτήστε το δικό σας το, το, το δικού σας εκλογής, του δικού σας ψηφοφόρους, αν θέλουν να γίνει μια τέτοια επανεγκατάσταση. Και θα δείτε για ποιο λόγο διστάζουν τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά το βόρειο κοσυφοπαίδιο. Το θετικό αν μπορώ να πω ότι είναι θετικό, είναι ότι ακόμα και τα κράτη, ε, τα, τα ε, δεν υπάρχει θέμα του κατά πόσον το βόρειο κωσυφοπέδιο ανοίξει το κωσυφοπέδιο, ακόμα και μεταξύ των χωρών που δεν αναγνωρίζουν την ανεξαρτησία του Ο Τώρα, ε, στην πράξη έχουμε σημαντικό πρόβλημα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. την ε, Άνοιξη ε, είδατε ότι και η αποστολή και το ΝΑΤΟ ε, έλαβαν μια πολύ αυστηρή στάση σε ό,τι αφορά τα συνορικά φυλάκια. Η πρόσβαση ε, της ε, πρόσβαση στο συνολικό φυλάκιο που ήταν να χρησιμοποιηθεί ε, μπλοκαρίστηκε και από την Κωσυφοπέδιο και από τη Σερβία και δεν χρησιμοποιήθηκε. Πρέπει να επιτύχουμε λοιπόν πρόοδο στο διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών. Παρόλο, τα, παρόλο το ότι είναι προβληματικός, το είπε και ο Φερνάντο Τζεντιλίν, πρέπει να προχωρήσει, πρέπει να εφαρμοστούν οι αποφάσεις, συμφωνίες. Εμείς είμαστε συγκρατημένοι αισιόδοξοι, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τα αποτελέσματα ασφαλώς. Ε, για το είπε Dick Marty, ε, μάλλον για την έκθεση του Dick Marty. Υπάρχει μια ερευνητική ομάδα ε, στο πλαίσιο της αποστολής. Οργανωτικά είναι σχετικά ανεξάρτητη από την αποστολή όμως. Συνεργάζεται με, την, με το δικαστικό σώμα του Κωσυφοπεδίου με αρκετές επιτυχίες σε ό,τι αφορά τη δημιουργία του απαραίτητου πλαισίου και συνεργάζεται και με το δικαστικό σύστημα άλλων κρατών και αναμένουμε ότι θα αρχίσουν οι επίσημες ε, δικαστικές έρευνες σύντομα σύμφωνα με το νόμο του Κωσυφοπεδίου που εφαρμόζεται θα έχει δύο χρόνια για να ολοκληρώσει το έργο της. Είναι μια σαφής προθεσμία. Μετά η υπόθεση θα πρέπει να προχωρήσει στην ακροματική της διαδικασία αν υπάρχουν ε, επαρκή πιστήρια και αποδεικτικά στοιχεία. Συλλήψεις στο βόρειο κοσυφοπαίδιο και η ε, δημοκρατική παρακολούθηση. Είναι δύσκολο να προβαίνουν σε ε, συλλήψει στο βόρειο κοσυφοπαίδιο. Μόλι συλλάβουμε κάποιον, βγαίνει όλο ο κόσμο στον δρόμο, φτιάχνουν οδοφράγματα, διαδηλώνουν και Μπορεί βέβαια να επιστρέψει κανείς ε, με τους ε, συλληφθέντες ε, στο υπόλοιπο κοσυφοπέδιο, αλλά μπορεί να θέσουμε έτσι κίνδυνο ζωές. Και το ερώτημα είναι αν έχουμε και επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Ξέρουμε ότι ο κ. Βυσελίνοβιτς, για παράδειγμα, είναι ένας εγκληματίας στο βόρειο κοσυφοπέδιο. Το θέμα είναι όμως έχουμε αρκετά στοιχεία, έχουμε αρκετούς μάρτυρες. Ε, έχουμε στοιχεία από το ε, ε, υλικά πιστήρια, από τη σκηνή του εγκλήματος, από τον τόπο του εγκλήματος. Ο κ. Βυσελίνοβιτς, όπως ξέρετε, στην περίπτωση οι Σέρβοι μάλιστα μας βοήθησαν. Την, τον συνάλαβαν οι ίδιοι στην επικράτεια του Βορείου, στο, στο έδαφος του, μάλλον στη δική τους επικράτεια. Νομίζω ότι απάντησα πολλά ερωτήματα. Σε ε, ό,τι αφορά την αντικατάσταση του επικεφαλής αποστολής. Υπάρχει ένα πρόβλημα στη διαδικασία επιλογής. Γνωρίζουμε ότι ο επικεφαλής θα ολοκληρώσει τη αιτία του. Δεν ξέρουμε όμως πότε ακριβώς. Μόνο αυτό μπορώ να σας πω. Όπως γνωρίζετε οι διαδικασία επιλογής είναι ε, διαδικασίες έτσι ε, απόρριτες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χάμπερ. Θα... Ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον επικεφαλή τη Αποστολή κύριο Μπούτι Μαρνάκ. Ευχαριστώ. Οι περισσότερε ερωτήσει καλύφθησαν από του προλαλήσαντε. Εγώ θα ήθελα μόνο να επικεντρωθώ σε ένα-δύο σημεία, για να απαντήσω να εξηγήσω ή να θυμίσω σε ποιο περιβάλλον ε, λειτουργούμε. Στις 15 Οκτωβρίου του 2010 ανέλαβα. Μέχρι τότε η αποστολή λειτουργούσε σε ένα περιβάλλον κρίσης. Και μπορώ να σας πω ότι και μέχρι τώρα είναι ένα ατέρμονο περιβάλλον κρίσης ο πρόεδρος ε, αναγκάστηκε να παραιτηθεί της χώρας. Εκολούθησαν εκλογές που δεν ήταν τόσο εύκολη υπόθεση. Ε, ε, χρειάστηκε μέχρι τον Απρίλιο για να ολοκληρωθούν το 2011 και πέρσι το καλοκαίρι, θυμάστε όλοι τι έγινε ελπίζω, το 10 Σεπτέμβριο επανήλθαμε σε μια κατάσταση πάρα πολύ τεταμένη. Και ο μόνος τρόπος να φτάσει κανείς στο βορρά στα σημεία εισόδου ήταν με ελικόπτερο για αντικατάσταση του προσωπικού. Ιδιαίτερα ένα σταθμό ο ένα καταστράφηκε ε, το καλοκαίρι και ε, ακολούθησαν εκλογές στη Σερβία και υπήρχε ανάγκη πώς να το πω, να κατευνάσουμε λίγο τις δραστηριότητές μας. Και αν είναι κανείς αρκετά ειλικρινής ε, για να παρακολουθήσει τι γίνεται, θα διαπιστώσει ότι ε, μόλις ε, ολοκληρώθηκαν οι εκλογές στη Σερβία πριν από μια μισή εβδομάδα, επαναλάβαμε ε, αμέσως τις αποστολές μας και στο Βόρειο Κοσφοπέδιο υπό πολύ δύσκολες συνθήκες κάναμε έρευνα σε καταστάσεις στο σπίτι του κυρίου Βερσίνοβιτς που όπως ξέρετε κρατείται στη Σερβία κάπου το τελευταίο διάστημα. Νοτίως του ποταμού Ήμπαρ γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα δίκτυο μεικτό διεθνές όπου συμμετέχουν ε, κακοποί και Αλβανοί και από το Βόρειο Κωσυφοπαίδιο. Όλα αυτά ε, συνιστούν λοιπόν ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργήσουμε. Υπάρχουν χώρε που αναγνωρίζουν, που δεν αναγνωρίζουν ζητήματα νόμου. Ε, αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Θα ήθελα να προσθέσω και κάτι για την εντολή μας. Η στρατηγική αναθεώρηση, νομίζω το είπα, ε, ορίζει ρητά ότι δεν υπάρχει αλλαγή στην εντολή. Υπάρχει αλλαγή στο κέντρο βάρους, αλλά η εντολή παραμένει ίδια. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν άλλαξε η κοινή δράση. Και νομίζω εκεί συμφωνούν όλα τα κράτη-μέλη να μην αλλάξει η κοινή δράση που καθορίζει και προσδιορίζει ε, την εντολή. Και ό,τι κάνουμε εμείς και ό,τι κάνω εγώ ιδιαίτερα συνδέεται με αυτό το κείμενο γιατί είναι ένα κείμενο ιδρυτικό που ορίζει ποια είναι η εντολή μας και τι αναμένεται από την αποστολή αφενός και αφετέρου. Εγώ κάνω αυτά που μου ζητούν και που μου έχουν αναθέσει τα κράτη-μέλη ε, από την ε, PSE και μην νομίζετε ότι ως επικεφαλής εγώ της αντιπροσωπείας κάνω κάτι διαφορετικό, οτιδήποτε διαφορετικό από το να ακολουθώ τους κανόνες. Σέβομαι την εντολή για την κοινή δράση αφενός και από την άλλη ακολουθώ τις εντολές που παίρνω από τα κράτη-μέλη. Ε, μέσω του PSE και η στρατηγική αναθεώρηση αυτό είναι. και ε, σας είπα ότι το περιβάλλον μεταβάλλεται και με ταχύς ρυθμούς. Και αυτή είναι η κατάσταση. Και σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη θα ήθελα να τονίσω και να επιμείνω ότι η κοινή δράση ορίζει ρητά ότι βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές εφαρμόζονται και προδιαγραφές. Οι ε, δικαστές είναι ανεξάρτητοι και αυτόνομος ο εισαγγελέα. Και μπορώ να σας πω ως ε, επικεφαλής αντιπροσωπείας προσέχω πάρα πολύ να σέβομαι αυτές τις βασικές αρχές ε, γιατί είναι απλές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φαντάζομαι κανείς εδώ δεν αναμένει τίποτα διαφορετικό από μένα παρατηρώ με ευλάβεια αυτές ε, τις ε, αρχές. Ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Μωρίνα. Ο κύριος Πόσελτ. Ζητώ συγγνώμη. Εγώ ρώτησα τι δυνατότητες καταγγελίας και παραπώνων έχει κάποιος. Κύριε Ντεμανιάκ, αυτό που σας ρώτησα εγώ ήταν ποιος μπορεί να κάνει παράπονα και καταγγελία στην ε, Γιούλεξ και μέσω της Γιούλεξ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τους πολίτες και θέλω να μου απαντήσετε. Μπορείτε να δώσετε τέτοια απάντηση. Υπάρχει ένας μηχανισμός για να γίνεται αυτό ένας ανεξάρτητος μηχανισμός, ο οποίος δεν είναι αυστηρά τμήμα του Γιούλεξ, αλλά συνεργάζεται στενά με τη Γιούλεξ και ε, λαμβάνουμε διαμαρτυρίες. Δεν έχω τώρα τα στοιχεία δυστυχώς, αλλά αναμηνία βάση υπάρχει μια έκθεση και βλέπουμε τι γίνεται με αυτές τις αγωγές. Κάποιες από αυτές... Ε, ε, δεν ε, προχωρούν διότι από νομική σκοπιά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να τις κλείσουμε αλλά ε, πολλές από αυτές τις διαχειριζόμαστε με τον κατάλληλο τρόπο υπάρχουν αναφορές σε τακτική βάση και εξηγούμε αναλυτικά τι γίνεται με όλα αυτά τα θέματα. Ε, ναι, υπάρχει λοιπόν μια διαδικασία και λαμβάνουμε υπόψη όλες αυτές τις διαμαρτυρίες. Ωραία, νομίζω ότι είναι πιο σαφή τα πράγματα. Η κυρία Μωρίνα τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω η ερώτηση για μένα ήταν κατά πόσον είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε εμεί ε, τα ημεία εγώ εξορισμού πιστεύω ε, ε, στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Δεν είναι θέμα του κατά πόσον είμαστε διατεθειμένοι ή μη να το κάνουμε. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Ε, πρέπει να είχαμε αναλάβει στις 18 Φεβρουαρίου του 2008 την κατάσταση, αλλά δεν έγινε για διάφορους λόγους. Το Κωσυφοπαίδιο είναι μια ανεξάρτητη χώρα, θα πρέπει να γίνεστε σεβαστό ως ανεξάρτητη χώρα και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο στο πολιτικό τοπίο που έχουμε στο Κωσυφοπέδιο αυτή τη στιγμή, ή μάλλον η απεικόνηση του το πολιτικού τοπίου, είναι αποτέλεσμα 23 ετών ε, πολύ δύσκολων ε, περιόδων του Κωσυφοπεδίου. Δεν νομίζω ότι είναι η πραγματική εικόνα όμως του Κωσόβου. Υπάρχουν δυνατότητες, αλλά οι δυνατότητες αυτές ε, δεν είναι αυτή τη στιγμή έτοιμες να ενταχθούν ε, στα των καιρών και νομίζω ότι ε, τα όσα γίνονται αυτή τη στιγμή μας βοηθούν να κρατήσουμε αυτή την εικόνα σε αυτή την κατάσταση. Ε, τι γίνεται, εάν δεν πάει καλά η εκλογική διαδικασία μπορούμε να έχουμε τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο μας στήριξε μεν αλλά υπήρχε και μια άλλη δήλωση λανθασμένη ε, δήλωση μάλλον ε, λέγοντας ότι η διαδικασία ήταν δημοκρατική και ελεύθερη. Δεν ήταν αλήθεια. Υπήρχαν πολλά λάθη και τελικώς καταλήξαμε με το ίδιο πολιτικό τοπίο που είχαμε και τα τελευταία χρόνια. Ειλικρινά λοιπόν ο χώρος για άλλες εναλλακτικέ λύσεις για να μπορέσουν να έρθουν στην επιφάνεια οι δικές μας η δυνατότητα και να οδηγηθεί η διαδικασία προς τη σωστή κατεύθυνση δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί και ίσως εδώ είναι που χρειαζόμαστε και τη βοήθεια των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μωρίνα. Και τέλος να δώσω το λόγο και στον κύριο Χούν. Να ξεκινήσω με μια προσωπική παρατήρηση ότι αφορά τη δημοφιλία της Γιούλεξ. Ίσως αυτό σχετίζεται και με την αποστολή της Γιούλεξ. Ε, το... Είναι προφανές ότι ο κόσμος ε, δεν θέλει κάποιον ε, να επιτηρεί την ανεξαρτησία και ο κόσμος είναι ανυπόμονος και αυτή η ανυπομονησία μεταφέρεται και βαρύνει την Γιούλεξ. Όμως αυτό πρέπει να γίνει. Η εισηγήτρια ρώτησε πού θέλουμε να είμαστε μετά από δύο χρόνια. Ποιο είναι το όραμά μας. Μια διαδικασία συγκριτικής ε, ανάλυσης έχει ήδη ξεκινήσει και οι στόχοι καταγράφονται σε αυτή τη διαδικασία. Για παράδειγμα, ε, θέλουμε ε, προ, προ, πρόοδο προς ένα πολυεθνικό σύστημα δικαιοσύνης, τελωνιακές ε, υπηρεσίες χωρίς παρεμβάσεις από πολιτικούς μέσα σε ένα υγιές πλαίσιο, συντονισμός και συνεργασία με όλα τα μέρη, ε, διεθνείς προδιαγραφές, προκειμένου να ε, προσφέρονται υπηρεσίε ε, που θα ανταποκρίνουν τι ανάγκε τη κοινωνίας χωρίς ε, διεθνές, διεθνείς παρεμβάσεις ή υποκατάσταση. η δεδηλωμένη στόχη. Θα χρειαστούμε χρόνο. Πόσο χρόνο. Δεν ξέρουμε πόσο χρόνο. Θεωρίζουμε την αποστολή μας με βάση τους στόχους μας. και πάλι να αναφερθώ στην στρατηγική αναθεώρηση, γιατί επικρίθηκε από κάποιους. Ε, ίσως ε, δεν έχω, ε, λένε ότι δεν έχουμε αντιμετωπίσει εστιασμένα τα κρίσιμα σημεία. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Ένας από τους στόχους της αναθεώρησης είναι η ανακατανομή του, του ανθρώπινου δυναμικού και των πόρων. Και αυτό γίνεται η Κομισιόν ε, έχει ε, προβαίνει σε ένα του, του, πληθυσμού, του προσωπικού. Ίσως ε, θα μπορούσαμε να πάρουμε κάποιο προσωπικό από την καθοδήγηση των μέτρων και να το περάσουμε σε άλλες δραστηριότητε, για παράδειγμα στο δικαστικό τομέα, γιατί εκεί έχουμε πολλή δουλειά. Επίσης, ας σκεφτούμε αν μπορούμε να μεταφέρουμε ανθρώπινο προσωπικό στο βορρά γιατί η Γιόλεξ πρέπει να εξασφαλίσει ψηλή ο, παρουσία, μάλλον με, ε, ισχύρη παρουσία και στο βορρά. Χρειάζεται να απελευθερώσουμε ε, επίσης ε, πόρους προκειμένου να κάνουμε και εξοικονόμηση ε, κονδυλίων. Ε, μιλάμε για μια μείωση του προσωπικού κατά 25%. Το ζήτησαν τα κράτη-μέλη και πρέπει να κάνουμε εξοικονομήσει κι εμείς. Συνεπώς, βάλαμε τα θεμέλια μέσω τη στρατηγική αναθεώρησης και η οποία θα πρέπει τώρα να γίνει πράξη. much, Mr. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χούν. Θα ήθελα τώρα να ευχαριστήσω κλείνοντα όλου του προσκεκλημένους για την ακρόαση. Νομίζω ότι μάθαμε περισσότερα. Μας, είδα, ε, μας παρουσιάσετε τις απόψεις σας ε, εκ των έσω. Σας ευχαριστώ πολύ και προσβλέπουμε να σας ξαναδούμε στην Επιτροπή μας. Να περάσουμε κατευθείαν στο επόμενο σημείο, αλλά πριν περάσουμε στο επόμενο σημείο θα ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση για την προηγούμενη έκθεση. Την έκθεση του κυρίου Μπρόκ για την ΚΕΠΑ, Κοινή Εξωτερική Πολιτική Ασφάλεια και Άμυνα, ε, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 27 Ιουνίου στι 12 το μεσημέρι. Ε, συζήτηση τη Δευτέρα 2 Ιουλίου στη Στρασβούργο και ε, η ψηφοφορία και πάλι στις 5 Ιουλίου στο Στρασβούργο. Αυτό για την έκθεση για την ΚΕΠΑ. Και τώρα, συνάδελφοι, να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Λίγο ησυχία, παρακαλώ. The next point Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η ενημέρωση από τον κύριο Παντζέρη ε, σχετικά με την κοινή επίσκεψη τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, τη Επιτροπή Προπολογισμών και τη Αντιπροσωπεία για τη σχέση με τι χώρε του Μαγκρέμ στην Τινησία από 2-5 Απριλίου του 2012. Ο κύριος Παντσέρη απέστειλε μια επιστολή για αυτή την ε, κοινή αποστολή. Η επιστολή έχει διανεμηθεί σε όλα τα μέλη της Επιτροπής και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ήταν τρει οι στόχοι αυτή της κοινή αποστολής να αξιολογήσει ποια κατάσταση βρίσκεται η πολιτική μετάβαση και η σταθερότητα του νέου καθεστώτο στην Τινησία ε, να δούμε τι επιχειρησιακέ ανάγκε τη Τινησιακή κυβέρνηση και να δούμε κατά πόσον ε, χρησιμοποιούνται καταλήλω τα ευρωπαϊκά ταμεία ε, συνεργασία. Να σα πω επίση ότι στι 4 Ιουνίου θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων εδώ στην Επιτροπή μα με τον Μουσταφά Μπεν Γιασάφ, ε, επικεφαλής της ε, συντακτικής συνέλευσης για τη ε, διαδικασία της μετάβασης στην Τινησία. Κύριε Παντζέρη, να σας δώσω το λόγο ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Καταρχάς, να ευχαριστήσω από πλευρά για τη βοήθεια που μας προσέφερε η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη Δινησία, Μας βοήθησε στη διάρκεια όλης αυτής της αποστολής. Να σας υπενθυμίσω ότι ήταν μια κοινή αποστολή ε, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Προϋπολογισμών και Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ. Οι στόχοι ήδη αναφέρθηκαν από εσάς, ε, δεν χρειάζεται να τα ξαναπώ εγώ. Όπως ε, θα είδατε και από το πρόγραμμα, η αποστολή αυτή ήταν μια ευκαιρία να επισκεφθούμε κάποια προγράμματα τα οποία χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνουν κάποιε συναντήσει υψηλού επίπεδου με τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία τη Τινησία, ε, τον Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων, τον Υπουργό Οικονομικών, ε, Περιφερειακές Ανάπτυξης, Διεθνούς Συνεργασίας και αρκετέ οργανώσει ε, και επιχειρηματιών και συνδικαλιστικές οργανώσει, και εκπροσώπους τη Κοινωνία των πολιτών, καθώ επίση και εκπροσώπου των ε, ε, κυριαρχών πολιτικών κομμάτων. Πρέπει να πω ότι καλό θα ήταν να ζητήσουμε και από την Επιτροπή Προϋπολογισμών να γίνει και μια επαλήθευση των ε, στοιχείων που δόθηκαν για την ε, χρηματοδότηση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην την Ισία. Είχαμε και μια ευκαιρία για να κάνουμε την πρώτη διμερή συνάντηση με τα μέλη της συντακτικής συνέλευσης. Θα ήθελα να καλωσορίσω και δύο μέλη της συντακτικής συνέλευσης Μπέικιν Φάι και Μπελκασιέν, οι οποίοι είναι εδώ για τη σημερινή συνεδρίαση. Η παρουσίαση τους εδώ αποτελεί ένα πρώτο βήμα ε, για μια στενή κοινοβουλευτική συνεργασία Στη διάρκεια αυτή της συνάντησης που είχαμε με τη συντακτική συνέλευση συζητήσαμε και το θέμα της στήριξη που δίνεται στη συντακτική συνέλευση και σε πολιτικό αλλά και σε διοικητικό επίπεδο και στη συνέχεια αυτής της ε, συνάντησης διοργανώθηκε μία ε, παραμονή μελέτης, διαμονή μελέτης για κάποια μέλη εδώ στις Βρυξέλλες ε, κάποιες πολιτικές σκέψεις. Είναι προφανές και από τα όσα είδαμε σε αυτή την αποστολή ότι η δημοκρατία σε αυτές τις αραβικές χώρες είναι μια μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη και σε αυτή την περίπτωση και η συντακτική συνέλευση και η μελλοντική ε, συνέλευση της Τινησίας θα πρέπει να λάβει υπόψη ε, τα στοιχεία αυτά και θα χρειαστεί και μια μόνιμη υποστήριξη που θα τις επιτρέψει να δημιουργήσει κοινοβουλευτικέ δομές ε, που θα χαίρουν πολυφωνίας και σε θεσμικό αλλά και εθνικό επίπεδο. Επίσης θα πρέπει να επισημάνουμε ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αισιοδοξία στην Τινησία, κυρίως ε, σε σχέση με τη κατάσταση των άλλων χωρών της Μεσογείου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σταθεί και στο ύψος των προκλήσεων που δημιουργούνται, κυρίως των οικονομικών προσκλήσεων για να αντιποκριθεί και στι ανησυχίε ε, των Τινησίων να σας πω ότι η δημοκρατία στην Τινησία και στην όλη περιοχή σίγουρα θα είναι πολύ πιο ε, σταθερή εάν μπορούν να δοθούν και κάποιες οθήσεις σε θέματα ανάπτυξης και να δοθεί και μια εγγύηση για ένα μέλλον στις ε, ε, νέες γενναίες. Θεωρώ ότι είναι ανησυχητικά τα όσα ακούσαμε από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ε, του κ. Βίβο, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα ε, στο Στρασβούργο μας είπε ότι το 2012 και το 2013 θα είναι κρίσιμα χρόνια και οι πληρωμές ε, προς αυτές τις χώρες ε, θα είναι αντίστοιχες στις χρηματοπιστωτικές θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν υποστήριξη και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωση και αυτό είναι θέμα μεριστής διατάξεως. Θα πρέπει να υπάρξει επανακεφαλαίωση τη ε, επανακεφαλαιοποίηση ε, και εμείς δεν μπορούμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην ε, εξετάσουμε το ζήτημα αυτό. Το να δημιουργηθεί το κράτος ε, δικαίου ε, είναι κάτι σημαντικό, αλλά θα πρέπει να γίνει και μια σημαντική δέσμευση για την καταπολέμηση ε, των εγκλημάτων που διαπράττονται και να διασκεδάσουμε αυτή την ανησυχία που υπάρχει για αυτή την ατιμερουσία που πιστεύετε ότι υπάρχει. Θα πρέπει να το εξετάσουμε πολύ προσεκτικά το ζήτημα αυτό και να το εξετάσουν όλοι όσοι συμμετέχουν και στη συντακτική συνέλευση αλλά και εμείς. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, ότι θα ε, είναι εδώ ο πρόεδρος της συντακτικής συνέδελφης στις 4 Ιουνίου και θα είναι μια σημαντική ευκαιρία για να συζητήσουμε και να δούμε τι μελιγενέστε με την Τινησία. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Mr. for your... Ευχαριστώ κύριε Παντσέρη για την έκθεσή σας. Κανείς δεν έχει ζητήσει το λόγο από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα. Οπότε ας καλωσορίσω τον εκ, τους εκπροσώπους της ε, οποίες στην Ισία, στην Επιτροπή μας. Να δώσω το λόγο το, στον κύριο Χάιτεν Πέλγα Κέτσεμ, πρόεδρο του Κογκρέπου Πουλα είναι πολιτική ομάδα ε, στο Κοινοβούλιο της Τινησίας. Ε, θα μπορούσατε να μοιραστείτε τις σκέψεις σας μαζί μας. Ποιος παίρνει το λόγο? Καλώς ήρθατε. Μπεσριφά Αλή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ομιλία σας. Θα σας υπενθυμίσω τι έγινε στην Τινησία. Είχαμε εκλογές διαφανείς, απόλυτος διαφανείς. Όλοι το αναγνώρισαν. Έχουμε το πρόβλημα της ασφάλειας αυτή τη στιγμή ορισμένα μέσα μας ενημέρωση ε, το μεγαλοποιούν. Η Τινησία έχει ως στόχο να μην χρησιμοποιήσει τη βία έναντι των ακραίων στοιχείων που υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή μόνο διαπραγματευόμαστε γιατί δεν θέλουμε να επιστρέψουμε στο παρελθόν. Δεν θέλουμε να ε, γίνουμε όπως το παλιό καθεστώς. Όμω, τα εξτρεμιστικά στοιχεία είναι μειοψηφία, δεν αποτελούν κίνδυνο. Από πλευράς οικονομία τώρα. Ήρθαμε εδώ για να σας ζητήσουμε να ε, ενθαρρύνετε τις, ε, τους επενδυτές να έρθουν στην Τινησία. Τους περιμένουμε, θα τους καλωσορίσουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλούς ανθρώπους, πολίτες μας που φεύγουν, προσπαθούν να μεταναστεύσουν με ε, απίστευτα μέσα, με κίνδυνο τη ζωή τους. Δεν θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Θέλουμε να, ε, ε, έρθει, να έρθουν Ευρωπαίοι πολίτες ως τουρίστες, ως επιχειρηματίες για να μας βοηθήσουν να λύσουμε τα προβλήματά μας και για να, και για να πετύχουμε τη μεταπολίτευσή μας. Δημιουργήσαμε το Υπουργείο Δημοκρατικής Μετάβασης που θα προσπαθήσει να λύσει ακριβώς ορισμένα προβλήματα μεταξύ αυτών το θέμα των επιχειρηματιών που είχαν συνεργαστεί με το παλιό καθεστώς. Σας ζητώ μια ακόμα φορά ευγενικά να προσπαθήσετε να μας βοηθήσετε ε, απελευθερώνοντας ε, υπέρ του σημερινού καθεστώτος τα περιουσιακά στοιχεία του προηγούμενου καθεστώτος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και πάλι για τα καλά σας λόγια. και την άποψή σας ότι είναι σταθερή την Ισία και οι ακραίες εξεμιστικές δυνάμεις είναι περιορισμένες και δεν απειλούν τη μετάβαση στη δημοκρατία. Δεν ξέρω αν θέλω ο κύριος Παντζέρη να πει δύο λόγια για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Solo per dire questo, Ένα να πω. την Τινησία και θεωρούμε ότι αποτελεί πραγματικά εργαστήριο της ε, Αραβικής Άνοιξης και είναι η χώρα που ε, πρώτη από όλες τις υπόλοιπες ε, ξεκινά να ακολουθεί το δρόμο της δημοκρατίας και το έχει επιλέξει αυτό ο λαός της Τινησίας. Αφενός λοιπόν πρέπει να συνεισφέρουμε στα όσα μας ζητούν, πρέπει να ικανοποιούμε τα αιτήματα της Τινησίας, τουλάχιστον από οικονομική σκοπιά, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν δυσκολίες αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη, αλλά και για ένα ουσιαστικό στοιχείο της ε, οικονομίας της Τινησίας, τον τουρισμό. Ε, σαφώς και περιμένουμε πάρα πολλά από αυτή τη συντακτική συνέλευση και ελπίζουμε ότι κατά την... Ε, δημιουργία του συντάγματο της Τινησία θα ληφθούν υπόψη όλες οι αρχές της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων των ανθρώπων, της προστασίας ε, της ελευθεροτυπίας ε, και ούτω ε, Ελπίζω ότι αυτός θα είναι ο στόχος όλων, ώστε η Τινησία να γίνει πραγματικά σημείο αναφοράς όλης της περιοχή της Μεσογείου. Thank you very much, uh, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πανσέρη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, και την αντιπροσωπεία της στην Ισίας Εξονόματος της Επιτροπής μας. Σας εύχομαι ε, ό,τι επιθυμείτε και ε, καλή, δημοκρα... καλή μετάβαση στο δημοκρατία. Τελειώνει αυτό το θέμα και προχωρούμε στο επόμενο δημιουργία ενό χρηματοδοτικού μηχανισμού για την προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο. Είναι το τελευταίο μέσο χρηματοδότησης από τα έξι που συζητούμε στην Επιτροπή μας. Η συγγετής και για αυτό το θέμα είναι ο κύριος Λάμστορφ, ο οποίος παρευρίσκεται και το δίνω μέσω στο λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. I'll do in English, though, so everybody can understand. Θα τα πω αγγλικά για να καταλαβαίνετε όλοι χωρίς ερμηνεία. Λοιπόν, σχέδιο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μελέτη αντικτύπου ε, με πιστικό τρόπο αντανακλά ε, τη ισχυρά σημεία και τις αδυναμίες του μηχανισμού μέχρι σήμερα και είναι το νέο σχέδιο ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και αλλού είχαμε συζητήσεις και διαβουλεύσεις με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και άλλους και καταρτήσαμε την έκθεσή μας βάσει των αποτελεσμάτων αυτών των ε, συζητήσεων. Κάναμε πολλές τροπολογίες και θα σας εξηγήσω το σκεπτικό. Νομίζω ότι η βασική αρχή είναι είτε ανεξαρτησία από τις ε, αρχές των τρίτων χωρών και έχει ε, μια πραγματική αυθεντικότητα σε σχέση με τα άλλα προγράμματα και μέσα περιφερειακής συνεργασίας. Είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε σε θέματα ε, που δεν καλύπτονται από τα άλλα μέσα. Να σας πω δύο λόγια για αυτό το κείμενο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και να είναι ε, στεναρή και πρέπει για τα βασανιστήρια, τη θανατική ποινή, ε, τη κακοποίηση γυναικών, παιδιών κλπ. Στο διάλογο με τις χώρες αυτές οι ευρωπαϊκές αξίες θα πρέπει να προάγονται και μέσω άλλων ε, μηχανισμών. Τούτος ο μηχανισμός είναι συμπληρωματικός και δεν θα πρέπει να θεωρείται πρόφαση και δεν θα πρέπει να ε, παραγωνίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε ό,τι αφορά όλα τα άλλα επιμέρους θέματα, αναφέρονται στο άρθρο 2, στο πεδίο εφαρμογή. Θα ήθελα όμως να πω ότι ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός. Ε, θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να δοθεί βοήθεια από αυτό το χρηματοδοτικό μηχανισμό, να είναι προστιθέμενη αξία και συνεργασία. Και για να υπάρχει αυτή η συμπληρωματικότητα, το λέω και στην έκθεσή μου, χρειάζεται ε, μεγάλος βαθμός ε, συντονισμού και θα δείτε ότι το τονίζω πάρα πολύ στην έκθεση αυτό. Επίσης ε, και σε σχέση με τη δουλειά που έγινε στους άλλους μηχανισμούς χρηματοδότησης θα πρέπει να πούμε ότι η στρατηγική που ε, υλοποιείται τώρα για τον προγραμματισμό και τη γενική θέση του Κοινοβουλίου για το οριζόντιο μέσο για να συνάδει αυτό, προτείνω η ε, κατεξουδότηση πράξη να μπαίνουν στα έγγραφα στρατηγική και στον κανονισμό αυτό. Βάλαμε μια παράγραφο που αφορά τη συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Για μα είναι πολύ σημαντική αυτή. Θέλουμε να ε, είναι επιλέξιμα αν χρειάζεται για χρηματοδότηση για τα κοινοβούλια. Ε, βέβαια, ε, θα πρέπει να το δούμε όπω και με τα άλλα χρηματοδοτικά μέσα, εάν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτό το πεδίο. Αυτό συνάδει με τις συστάσεις του Κοινοβουλίου για την υποστήριξη της δημοκρατίας και λαμβάνει πλήρως υπόψη το πλήρω εκλογικό κύκλο, δηλαδή να μην πηγαίνουμε επιμέρους μόνο αποσπασματικά σε παρατήρηση εκλογών. Θα πρέπει να δίδεται συνέχεια σε αυτές τις αποστολές. Και ξέρετε ότι χρηματοδοτείται από το μηχανισμό αυτό και η παρατήρηση εκλογών. Επίσης, να χρησιμοποιήσουμε ε, κάποια άρθρα να τα βγάλουμε από το οριζόντιο έγγραφο και να τα εντάξουμε στο συγκεκριμένο μέσο, γιατί αυτό είναι το χρηματοδοτικό μέσο για τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις ε, διαδικασίες και σε αυτό τον κανονισμό ανήκουν αυτά. Ε, μερικές ειδικέ τροπολογίες αφορούν την επιχειρησιακή πλευρά και θα ήθελα να τονίσω ότι η αναθεώρηση του χρηματοδοτικού μηχανισμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία αφορά τη λειτουργία του. Το κείμενο είναι ξέρετε, τεχνικό και νομοθετικό και αρκετά στενό ε, το περιθώριο αλλαγών. Εμείς θέλουμε να υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη νέα έμφαση, ε, περισσότερη δυνατότητα αντίδρασης και άμεσης δράσης σε επίγουσες καταστάσεις με βοήθεια Δηλαδή να μην υπάρχει διαδικασία και ε, καμιά φορά άμεση ανάθεση και όχι να περνάμε από πρόσκληση, εκδήλωση ενδιαφέροντος για διαγωνισμούς όταν είναι επίγουσα κατάσταση. Η κοινωνία των πολιτών μας επικρίνει ότι δεν επωφελούνται λόγω της περιπλοκότητας του μηχανισμού πολλές οργανώσεις πολιτών επιτόπου, μικρές. Τα μεγάλα έργα έχουν πάρει από 600.000 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Γειτονία, ενώ υπάρχουν πολλοί ε, βέβαια μεγάλες ΜΚΟ που είναι πολύ επαγγελματικέ και μπορούν ε, να απορροφούν τέτοια κονδύλια, αλλά μικρές οργανώσεις ε, πολιτών μη κυβερνητικέ είναι τόσο μικρές και δεν μπορούν να απορροφούν τόσα κονδύλια. Γι' αυτό θέλουμε να υπάρχει δυνατότητα χορήγηση βοήθεια μέχρι 100.000 ευρώ με απλουστευμένη διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμών και να υποστηρίζονται οι οργανώσει στη λειτουργία και στη δομή του και σε κεντρικό επίπεδο, α πούμε από εδώ της Βρυξέλλη, και όχι μόνο ε, επιτόπου στις ε, δικαιούχε χώρε. Θα πρέπει να δούμε πώ αυτό θα ενταχθεί στο δημοσιονομικό κανονισμό, δηλαδή πώ μπορεί να γίνει συμβατό, Πάντω, αδύνατο δεν νομίζω να είναι. Επίση, υποστηρίζω την ίδρυση μιας ομάδας εργασίας διοργανική που να ασχολείται με την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών ε, δεν μπορεί να γίνει, όπως σας είπα, σε αυτό το κείμενο που είναι τεχνικό, αλλά ανεξάρτητα και παράλληλα με την νομοθετική διαδικασία, πιστεύω ότι μπορούμε να συστήσουμε μια τέτοια ομάδα για να έχουν πρόσβαση πιο μικρές και πιο τοπικές ΜΚΟ σε αυτή την προσπάθεια και τη χρηματοδότηση. Ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει επίσης, εμείς ζητήσαμε να μειωθεί οροφή για τα έργα σε πολύ δύσκολες καταστάσεις χωρίς ε, προκήρυξη διαγωνισμού Δύο εκατομμύρια είναι σήμερα ε, το ποσό αυτό. Μου φαίνεται υπερβολικό. Δεν ξέρω αν υπάρχει καλύτερη εξήγηση που την αγνοώ. Αν θεωρήσουμε ότι ε, η διάρκεια του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 18 μήνο, θεωρήσαμε ότι αυτή η οροφή είναι πολύ ψηλή ε, δεδομένου του συνολικού όγκου της χρηματοδότησης. Θα πρέπει να υπάρχει ένας ταχύς μηχανισμός απόκριση σε χώρες μετάβαση ε, για να ενισχύονται ε, αξιόλογα έργα. Το είδαμε στην Αραβική Άνοιξη, δεν καταφέραμε να προωθήσουμε αυτή την προσπάθεια. Ένα τελευταίο έχει να κάνει ε, πάντα με το μηχανισμό αυτό. Πώς θα συνεργάζεται και με το Μελλοντικό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία και ποια θα είναι η διαφορά του. Τώρα ολοκληρώνεται την προσπάθεια για το Ίδρυμα για τη Δημοκρατία και θα εργάζεται σε τομείς που μπορεί να ε, μας προβληματίζουν και μας ανησυχούν να μην υπάρχουν επικαλύψεις με το χρηματοδοτικό μηχανισμό. Λοιπόν, να δούμε τι μπορεί, τι πρέπει να κάνει, τι δεν πρέπει να κάνει το Ίδρυμα και τι μπορεί, δεν πρέπει να κάνει ο χρηματοδοτικός μηχανισμός για να μην έχουμε επικαλύψεις και διπλή δουλειά και είναι και πάρα πολύ έντονη η εντολή της Επιτροπής μας προς εμένα για να αποφευθούν αυτές οι επικαλύψεις και η παράλληλη δράση. Αυτά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα να ε, περιγράψουμε σωστά το κάθε μηχανισμό και το Ίδρυμα να συνεργάζονται, να μην έχουν αντιπαλότητες και επικαλύψεις. Το Ίδρυμα για τη Δημοκρατία ε, εστιάζεται περισσότερο σε πολιτικά ζητήματα, ενώ ο χρηματοδοτικός μηχανισμός ε, αφορά περισσότερο την κοινωνία των πολιτών και όχι τόσο τα πολιτικά κόμματα. Καλά, αυτά θα το ξανασυζητήσουμε τις επόμενες εβδομάδες και μήνες για να δούμε πώς μπορούμε τον καλύτερο τρόπο να το ρυθμίσουμε. Ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω στην ανταλλαγή απόψε. Ευχαριστώ κύριε Λάμστορφ. Ευχαριστούμε για αυτή την πολύ καλή έκθεση. Ο λόγος καταρχήν στον κύριο Κούκαν. Thank Παίρνω το λόγο εκ μέρου τη κυρία Μακοβέη, που είναι σκιώδη εκ μέρου του, ε, για το ΕΛΚ και δεν μπόρεσε να είναι παρουσά. Καλωσορίζουμε την καινούργια πρόταση της Κομισιόν. Είναι πιο αποτελεσματική και εκφράζει την προσήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίω μέσω των οργανώσεων ε, της κοινωνίας των πολιτών σε τρίτες χώρες. Το μέσο αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο, θα επιτρέψει να δίδεται βοήθεια ανεξαρτήτως ε, της σύμφωνης νόμης ε, το, της κυβέρνησης των τρίτων χωρών και αυτό το διαφοροποιεί από άλλα μέσα. Ε, χρηματοδοτικά χρηματοδοτικά μέσα εξωτερικής πολιτικής. Ε, έχει, είναι ισορροπημένο, ε, ανάμεσα ε, στις, ε, στους στόχους του. Νομίζουμε ότι είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε τα, τους υποστηρικτές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ενδεχομένως μπορεί να υφίστανται Απειλέ ή εκφοβισμό από τρίτα μέρη. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τους συνδράμουμε με τρόπο που δεν θα θέτει σε κίνδυνο την ακαιρεότητά τους. Ο εισηγητής διέγραψε το ποσό το οποίο αναφέρεται ε, του 1 δισεκατομμυρίου 58 εκατομμυρίων ευρώ. Πιστεύουμε όμως ότι θα πρέπει να βάλουμε τουλάχιστον ένα ελάχιστο ε, προπολογισμό. Θα επανέλθουμε με λεπτομερείς τροπολογίες σε επόμενες μέρες. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Εκ μέρους του Σωμάτου Σοσιαλιστών, κ. Χόουιτ. Εκ μέρους της κυρίας Γκόμες, θέλω να ευχαριστήσω τον Αλεξάνδερ. Ε, συνεργάστηκε πολύ καλά μαζί μας για όλα αυτά τα θέματα και υποστηρίζω πολλά από όσα είπε. Δεν θα τα επαναλάβω. Νομίζω ότι θα εξασφαλίσουμε συνένεση. Ευχαριστώ, Αλεξάνδρ. Θέλω να καταγραφεί το εξή. Ε, υπάρχει ανάγκη να υπογραμμίσουμε την διαβούλευση με τις οργανώσεις ε, της κοινωνίας των πολιτών, με τις ε, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επιτόπου κλπ. κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προγραμματισμού δεν είναι μόνο εκτελεστικά όργανα αυτές οι οργανώσεις. Θέλουμε να ζητείτε η γνώμη τους για τις προτεραιότητές μας, για τον προγραμματισμό μας. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε στους συναδέλφους της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι οργανώσεις και οι πληροφορίες που θα μας δίνουν θα προωθούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγκαιρα κατά τη διάρκεια τη ε, διαδικασία προγραμματισμού. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το αποφασίσουμε τώρα, όταν μιλάμε για το ονομαστικό κείμενο, όχι αργότερα. Γιατί αργότερα θα δημιουργηθούν καυγάδε σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στι πληροφορίε. Είμαι σίγουρο ότι ο Αλεξάνδρας θα συμφωνήσει μαζί μου. Σήμερα θα πρέπει επίση να αρχίσουμε και το θέμα των πράξεων κατά εξοδότηση. Πολλοί από εμά έχουν περάσει πολλές νυχτερινές ώρες ε, να καυγαδίζουμε ε, για την ε, υλοποίηση των υποσχέσεων που μας είχαν δοθεί. Τώρα θα πρέπει να αποφύγουμε τέτοιου είδου καυγάδες στο μέλλον και θα πρέπει να απαιτήσουμε ήδη από τώρα να εφαρμοστούν οι κανόνε λογοδοσία. Ο Αλεξάνδρ α το δει προσεκτικά και εμεί θα συνεργαστούμε μαζί του έτσι ώστε και το πνεύμα και το γράμμα τη συμφωνία να ε, καταγραφεί στο κείμενο. Συμφωνούμε με τον Αλεξάνδρ για την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία. Η υπηρεσία εξωτερική δράση έχει καλές προθέσει. Όλοι έχουμε καλέ προθέσει. Όμω η αλήθεια είναι και το ξέρουν όσοι έχουν εμπλακεί με τα θέματα του μέσου ε, τα τελευταία χρόνια υπάρχει ε, κίνδυνος για ε, ε επικίνδυνες δραστηριότητε των ανθρώπων που διαχειρίζονται το πρόγραμμα. Φοβούμε ότι πολλές φορές θα υπάρχει ο κίνδυνος αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη να μην είναι αυτοί που θα παίρνουν τα κονδύλια. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να ε, αναλάβει τους κινδύνους και ήδη η διατύπωση θα πρέπει να είναι τέτοια έτσι ώστε να το επιτρέπει αυτό στην Κομισιόν και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Σε πολλές περιπτώσεις άνθρωποι που δρούν με λιγότερο ορατό τρόπο επειδή φοβούνται για τη ζωή τους δεν πρόκειται να υποβάλουν επισήμω αιτήματα και αιτήσει για χρηματοδότηση κλπ. Ε, γνωρίζω τη θέση της Κομισιόν αλλά γνωρίζουμε επίσης και την πραγματικότητα. Συμφωνώ επίσης με την ανάγκη να δούμε πώς θα διαρθρωθεί ε, το μέσο αυτό με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία. Η κυρία Γκόμες θέλει να υποστηρίξει το έργο του Αλεξάνδρ και πάντοτε λέμε ότι το μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου ε, δεν θα πρέπει να περιθωριοποιήσει τις δαπάνες σε θέματα των δικαιωμάτων μέσω άλλων προγραμμάτων ή μέσων. Έχουμε ένα καινούριο μέσο, το ε, Ίδρυμα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και δεν θα πρέπει το ένα να ε, βάζει το άλλο στο περιθώριο, να επισκιάζει το άλλο. Σε ό,τι αφορά τι ε, αποστολές παρατηρητών, το έχουμε πει επανειλημμένως ότι αποτυγχάνουμε όχι στι αποστολές παρατηρητών, αλλά το, στο πριν και στο μετά. Θέλουμε όλο αυτό να είναι μια αλυσίδα μετάβαση στη δημοκρατία. Και εκεί είναι που ε, από την Ας βελτιώσουμε λίγο το κείμενο. Συμφωνώ επίσης με το, αυτό που είπε ο κύριος Κούκαν και ο κύριος Λάμστορφ ε, σε ό,τι αφορά το τι ποσό, τι ποσοστό μάλλον θα δαπανάτε σε κάθε δράση. Ε, ε, εντάξει να δαπανούμε για την παρατήρηση των εκλογών, αλλά να καθορίσουμε σωστά τα ποσοστά. Τώρα, ρόλος των ε, αντιπροσωπείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το μέσο για δημοκρατία και δικαίωμα, του ανθρώπου, επειδή ε, είχε μικρότερο ποσοστό χρηματοδότησης από ότι άλλα μέσα, ε, έχει χρησιμοποιηθεί πολύ καλά από και χειρότερα από άλλους. Το έχουμε δει αυτό σε αποστολές. Οπότε το μήνυμα προ την υπηρεσία εξωτερική δράση ε, πρέπει να είναι ότι όλε οι αντιπροσωπείε τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να συνδιαλέγονται με του δικαιούχου ε, τη χρηματοδότηση και να ενισχύουν τη δημιουργία τοπικών δυνατοτήτων έτσι ώστε να μπορεί να μπορούν οι οργανώσεις, μη κυβερνητικέ οργανώσει και οι οργανώσει κοινωνία των πολιτών να συμμετάσχουν. Και η διαφάνεια επίση είναι πολύ σημαντική. Η διαφάνεια δεν είναι μόνο, δεν σημαίνει ότι μόνο εμείς έχουμε πρόσβαση στα έγγραφα. Αν θέλουμε οι οργανώσεις, οι μη κοινωνικές οργανώσεις να ε, παίξουν σημαντικό ρόλο, θα πρέπει και αυτές να ενημερώνονται, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα στρατηγικής, να τα σχολιάζουν και να συμμετέχουν στην διαδικασία διατύπωσής τους. Οπότε το θέμα της πρόσβασης δεν αφορά μόνο τους ευρωβουλευτές αλλά και την κοινωνία των πολιτών. Νομίζω ότι αυτά είναι ανησυχίε κοινέ στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χαουτ. Δεν έχει ζητήσει άλλος το λόγο. Θα παρακαλούσα τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να μας πούν τις απόψεις Πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλημέρα σας. Ε, είμαι αναπληρωτής ε, ε, τμήματάρχης της μονάδας που ασχολείται με αυτό το θέμα. Δύο γενικά σχόλια. Βεβαίως να συγχαρούμε τον εισηγητή και όλους όσοι εργάστηκαν στην έκθεση αυτή. Για το θέμα συζητούμε με τα κράτη-μέλη και γιατί να μην συμφωνήσουμε στην πρώτη ανάγνωση επί της ουσίας του μέσου. Δεν μιλώ για τα θεσμικά ζητήματα, ούτε για τα δημοσιονομικά, τα οποία έχουν μεγάλες προεκτάσεις, αλλά σε ό,τι αφορά ε, τις συνομιλίες που είχαμε και την εξαιρετική κατεύθυνση που παίρνει αυτό το έγγραφο, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε επί της ουσίας πάρα πολύ γρήγορα. Δεύτερον, είπε και ο κύριος Λάμστορφ ότι μερικά από τα όσα πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόταση οριζόντιου κανονισμού ε, ανεβρίσκονται και εδώ. Δεν έχει σημασία ε, αυτό ε, που βρίσκονται αυτές οι διατάξεις αρκεί να μην είναι το ίδιο κείμενο ή αρκεί να μην είναι δύο διαφορετικές αναφορές σε διαφορετικά κείμενα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ουσία και όχι πολύ ο τύπος που θα ενταχθούν αυτά. Τα δημοσιονομικά συστήματα διαπερνούν όλες τις τροπολογίες που διαβάσαμε μεγάλο ενδιαφέρον και αφορούν γενικά όλα τα χρηματοδοτικά μέσα και δεν θα μπω στι λεπτομέρειε. Θα πω όμως κάτι για ε, το απόρριτο, για τη συμπροματικότητα και για την ευελιξία. Για το απόρριτο ή την εμπιστευτικότητα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να μοιραζόμαστε τις προφορίες, αλλά Χρειάζεται προσοχή γιατί υπάρχει ένα τμήμα του μέσου που είναι αρκετά περιοριστικό και θέλουμε να παραμείνει ε, αυτό επιστευτικό γιατί όταν δημοσιευθεί οποιαδήποτε πληροφορία ε, ε, απειλούνται οι ενδιαφερόμενοι. Θα πρέπει να ξαναδούμε τη διατύπωση. Βεβαίως οι βουλευτές να έχουν πρόσβαση αλλά ενδεχομένως όσοι το χρειάζονται, όχι και 700 τόσοι βουλευτές δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να το συζητήσουμε, να βρούμε έναν τρόπο να το διατυπώσουμε, να το ε, διαρθρώσουμε έτσι ώστε αυτό το εμπιστευτικό κομμάτι να παραμείνει εμπιστευτικό. Υπάρχουν και ε, πολίτες ε, δικοί μας ε, που είναι στη φυλακή επειδή δεν τηρήθηκε το απόρριτο. Συμπροματικό ναι, αλλά όχι δευτερεύον. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που συζητούμε, μπορεί και με άλλα ε, ε, ε, την υποστήριξη της κοινωνίας πολιτών, του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Δημοκρατία, το Endowment. Είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία, αλλά δεν είναι μόνη. Συμφωνώ με τα όσα ακούσαμε, όχι οι επικαλύψεις, αλλά κάτι πιο σημαντικό είναι η προσθετικότητα των κονδυλίων. Δηλαδή, είναι σημαντικό. Ανέκαθεν ακούμε ότι το Ίδρυμα θα περιορίζεται ε, στο ENPI και ότι τα κονδύλια αυτά θα ήταν επιπλέον. Να προσέξουμε τη διατύπωση και ε, να μην αντλήσουμε κονδύλια από το Ίδρυμα για τη Δημοκρατία, να βρεθούν επιπλέον κονδύλια από αλλού. Θέλει προσοχή αυτό. Και το τελευταίο για την ευελιξία. Δεν θα βρείτε ποτέ ε, υπάλληλο που να διαφωνήσει με την απλούστευση και τη βελτίωση της ευελιξίας. Οτιδήποτε τη βελτιώνει είναι ευπρόσδεκτο, αλλά θα πρέπει οι νομοθέτες να υπογράψουν την απλούστευση στην τροποποίηση ε, του ε, δημοσιονομικού κανονισμού που αυτό τον καιρό ε, είναι καθοδόν και έχει οδηγηθεί σε εμπλοκή στα νομοθετικά όργανα. Λοιπόν, ας υπογράψουμε πρώτα τις προτάσεις που έχουμε και μετά να ζητούμε νέες. Για τα νέα τώρα μέσα, κοινέ δυνατότητε. Ποια είναι η βασική καινοτομία στην πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακριβώ αυτή η δυνατότητα να υπερβαίνει κανεί ε, την ε, προκήρυξη διαγωνισμού σε χώρε που δεν έχει νόημα αυτή. Ε, λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα κατάργησης. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε για το κόστος. Ε, μικρές ε, βοήθειες είναι 50.000 ευρώ που έχουν χαμηλή προστιθέμενη αξία. Παράδειγμα, μπορέσαμε να δράσουμε στη Λιβύη σε μια κατάσταση κρίσης. Ε, δημιουργήσαμε ένα σύστημα περίθαλψης ιατρικής, ψυχιατρικής και επανένταξης πολλών εκατοντάδων γυναικών που είχαν υποστεί στη Λιβύη κάκο μεταχείριση σωματική και σεξουαλική. 1,5 εκατομμύριο σε 10 μήνες με 5.000 ευρώ ε, αντιμετωπίζουμε και 10 γυναίκες. Στη Λευκορωσία επίσης, επειδή έχει ξενθεί πολύ η κατάσταση, έχουν σκλίνει τα πράγματα και ε, ως προς τις ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μισό εκατομμύριο ε, μπορεί εκεί να αφιερωθεί νομική υποστήριξη. μπορούμε να βοηθήσουμε για ενημέρωση, εκπαίδευση πολιτικών κομμάτων στη Λιβύη, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ένα εκατομμύριο για 18 μήνες για να βοηθήσουμε τις γυναίκες να συμμετέχουν. Δηλαδή, 100.000 ευρώ να υπάρχει δυνατότητα αλλά 100.000 ευρώ τι σημαίνει, ότι βγάζουμε από την Κίνα 10, όχι 100 ε, ε, ε, αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά 100.000 ευρώ δεν αλλάζει και πολλά πράγματα στο σύστημα που ισχύει. Γι' αυτό ζητούμε να ε, φτάσουμε σε 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, ε, όπως είναι το μέσο σταθερότητας. Αυτό είναι η οροφή. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να εξαντληθεί, αλλά για να είμαι ειλικρινής, η οροφή 100.000 δεν αλλάζει πολλά πράγματα. Τώρα, για το θέμα των μικρών ε, δωρεών, μικρών ενισχύσεων, small grants, για 10.000 ευρώ μπορούμε να συγχρηματοδοτούμε μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Δηλαδή, είναι μεγάλη αλλαγή αυτό, ριζική αλλαγή προσέγγισης. Δεν ενισχύουμε οργανώσεις, ενισχύουμε δράσεις. Θα έχουμε κάποια προβλήματα ε, και για την προσέγγιση και για τα κριτήρια. Δηλαδή, σε ποια βάση μπορεί κάποιο να αρνηθεί σε μία ΜΚΟ χρηματοδότηση. Αν το δεχτούμε για όλε τι ΜΚΟ, θα πρέπει να το διαχειριζόμαστε με τον ίδιο τρόπο, ε, με ε, πακέτα 10.000 ευρώ κάθε φορά. Ανοίγει πολύ η πόρτα επίσης στις προσωπικές επιλογές και αυτό είναι πρόβλημα. Επίσης θα πρέπει να τριπλασιαστεί το κονδύλι το διοικητικό και ε, το στελεχειακό μας δυναμικό για να διαχειριζόμαστε τέτοια πακέτα των 10.000 ευρώ. Τώρα, επί της ουσίας, αυτό που λέμε τα μικροέργα, τα πολύ μικρά έργα. Να παραμείνει αυτό, η λογική μέχρι τώρα τι έλεγε να διαιρείται σε δύο τμήματα. Ε, το τμήμα που διαχειρίζεται μια αντιπροσωπεία που κάνει πραγματικά μικροέργα και ενώ η έδρα ε, τα κεντρικά ε, ασχολούνται με τα μεγάλα έργα. Είναι δύσκολες χώρες που έχουν μεγάλο κόστος και μεγάλοι φορείς και λόγω του μεγέθους έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα. Αν αλλάξει αυτό χρειάζεται πολλοί κόσμος για να το διαχειρίζεται. Και ένα τελευταίο να απαντήσω για δύο πράγματα. Για την Αραβική Άνοιξη. Δεν νομίζω ότι δεν κάναμε τίποτα. Ε, ίσα ίσα. Ε, είμαστε παρόντες ε, σε πολλές χώρες πριν την Αραβική Άνοιξη για να υποστηρίζουμε τις οργανώσεις που συχνά δραστηριοποιήθηκαν εκεί. Στην Τινησία είχαμε πάει πέντε μέρες μετά την πτώση του Μπεναλή σχετικά γρήγορα, ακόμα και από πριν το μέσο σταθερότητας. Είμαστε παρόντες σε όλες τις χώρες Αραβικής Άνοιξης και εντό δεκαπεθημέρου θα εκδώσουμε ένα έγγραφο γιατί μας προσάπτουν πολύ συχνά τι κάνατε στην Αραβική Άνοιξη ότι δεν κάναμε αρκετά επειδή δεν έχουμε αρκετά κονδύλια εντάξει αυτό μπορεί να ισχύει αλλά ότι κάναμε κάναμε ε, για το θέμα του λόγου της σχέσης ε, συμφωνώ αλλά να μην συζητάμε μόνο για ένα κλάσμα του μέσου. Ε, ε, ωραίες εκλογές, σημαντικές, αλλά όλα αυτά θα τα πρέπει να, να τα βλέπουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο γιατί τα κονδύλια είναι δεδομένα και όταν χρηματοδοτείς δεξιά δεν χρηματοδοτείς την αριστερά σου. Αν είναι κατεξοδότηση πράξη, έστω. να συμφωνήσουμε με ποιο τρόπο θα ε, κατανέμονται τα κονδύλια για να μην υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Αυτά. Είναι πολλά τα σχόλια και τεχνικά και θα επανέλθουμε. Μερικά στοιχεία συμβατότητα με το δημοσιονομικό κανονισμό που πρέπει να δούμε για τι προτάσει για τη συνυπευθυνότητα, το επίπεδο δηλαδή η χρηματοδότησης. Δεν μπορούμε να το καταργήσουμε τελειώ. Μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα αν θέλετε, αλλά υποστηρίζουμε όλε τι προτάσει. Και βεβαίω ενδιαφερόμαστε να συζητήσουμε σε μεγαλύτερε λεπτομέρειε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη ε, εμπεριστατωμένη παρέμβαση. Ο κύριος Χάουιτ. Μία ερώτηση στον κύριο Λάμστρομ. Κάτι επιπλέον σε απάντηση σε αυτό. Εγώ ποτέ δεν έχω ακούσει για παραβίαση της εμπιστευτικότητας ε, μέσω Ευρωβουλευτών ή του Κοινοβουλίου όταν συζητάμε αντίστοιχα θέματα στο παρελθόν. Δεν μας κατηγόρησε κανείς για κάτι τέτοιο είχε μείνει να πλανάται στον αέρα. Θα ήθελα να καταγραφεί αυτό και θα ήθελα να καταγραφεί επίσης ότι όσοι έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες ε, διατηρούν την εμπιστευτικότητα προς όφελος της ασφάλειας των ανθρώπων και δεν υπάρχει καμία διαφορά ε, μεταξύ ημών και οποιοδήποτε άλλου. Και θα ήθελα επίσης να πω υπάρχει διαρθρωμένος διάλογος ε, για τα θέματα αυτά όταν ε, συναντώμαστε ιδιαίτερος. Ε, δεν υπάρχει παραβίαση όπως είπε και ο κύριος Λάμστρουγκ αναφέρθηκε στο θέμα της απλούς φεστευσής και με βάση αυτά που ακούσαμε καλό θα ήταν να υπάρχει στο συγκεκριμένο ψήφισμα και ο διαρθρωμένος διάλογος. Το έθεσα το θέμα αυτό και στη Βαρονιά στην Ολομέλεια, το επιβεβαίωση Καλό θα ήταν λοιπόν να, γίνει, ε, να ληφθεί υπόψη για οποιαδήποτε νέα παρατήρηση ή παρουσίαση, να το αναφέρετε αυτό για το διαρθρωμένο διάλογο και δεν μην χρειάζεται να σας το υπενθυμίζουμε εμείς. Ε, θα είναι καλό για την τήρηση της εμπιστευτικότητας από όλες τις πλευρές. Ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο σας. Κάποιος από πλευράς Επιτροπής ή από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα ήθελε το λόγο να επανέλθω στο σημείο αυτό. Ποτέ δεν είπα ότι υπήρξε παραβίαση της εμπιστευτικότητας. Ε, είμαστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε, αλλά θέλουμε να επεκτείλουμε το σύστημα του απορρίτου και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το πώς θα το κάνουμε. Δεν λέμε ότι δεν πρέπει να γίνει. Εμείς δεν δίνουμε πληροφορίες ακόμα και σε άλλες ε, τμήματα της... Ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ούτε και σε όλα τα κρατημέλη. Όταν λέω ότι πρέπει να είναι διαρθρωμένα, ε, λέω ότι θα πρέπει να παραμείνει το πολύ καλό επίπεδο εμπιστευτικότητας. Εγώ ήθελα να πω εξαιρετική ιδέα μεν, αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν επιπλέον και να υπογραφούν πολύ γρήγορα. Για παράδειγμα, ο τρέχον δημοσιονομικό κανονισμό, ο οποίο ακόμα δεν έχει υπογραφεί. Ε, και έχουμε ανέβει από τα 100.000 ευρώ στα 500.000 ευρώ. Μπορούμε δηλαδή να πολλαπλασιάσουμε επί 5 ε, το, η βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε. Ξέρω πολύ καλά σε τι θέση βρίσκομαι. Απλώ λέω ότι επιπλέον αυτού θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και αυτή την ευκαιρία για να υπογράψουμε ό,τι μπορούμε να υπογράψουμε πολύ γρήγορα για να έχουμε και επιπλέον ευελιξία από αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Υπάρχει κάποιο άλλο από την υπηρεσία τη εξωτερική δράση, την Κομισιόν, που να θέλει να λάβει το λόγο. Όχι, ο Αλεξάνδρ, παρακαλώ. Σε ό,τι αφορά το σχόλιο του κ. Κούκαν, ε, έχει σχέση με τη γενικότερη συζήτηση για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Συμφωνώ μαζί του ότι ε, δεν το είχαμε προβλέψει. Δεν θα πρέπει ε, να παραβαίνουμε τις ε, δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει. Η Επιτροπή Προπολογισμών νομίζω δουλεύει για αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή. Πρόσβαση πληροφορίας εμπιστευτικότητα. Η ανταλλαγή απόψεων έδειξε ότι ε, είναι δυνατόν η Κομισιόν δείχνει δεκτικότητα, ε, μπορεί, θέλει να δουλέψει αυτό το θέμα. Σίγουρα κάποιες πληροφορίες πρέπει να ε, είναι εμπιστευτικές με περιορισμένη πρόσβαση το επιτάσσει η φύση των πληροφοριών αυτών. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε μια λύση. Ευχαριστώ για την ευκρίνηση. Δεν υπάρχει μέχρι τώρα κανένα είδου παράβαση τη αρχή εμπιστευτικότητα στο παρελθόν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σημαντική διαφωνία ούτε ανάμεσα στι πολιτικέ ομάδε, ούτε ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την Κομισιόν. Το ίδιο και για την ευελιξία. Και εδώ νομίζω έχουμε συνένεση άκουσα τους συναδέλφους και τον Πατρίς, το θέμα από ό,τι καταλαβαίνω είναι το εξής. Θα πρέπει όπως πρότεινα εγώ να έχουμε μια παράλληλη ομάδα εργασίας, παράλληλη δηλαδή με την νομοθετική διαδικασία ή όπως πρότεινε εσύ να ε, συμπεριλάβουμε τον ε, διαρθρωμένο διάλογο εντός της ε, δια, ε, νομοθετικής διαδικασίας. Αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε. Επί της ουσίας όμως δεν βλέπω κανένα πρόσκομα. για το ρόλο των αποστολών παρατηρητών εκλογών. Ε, όλοι συμφωνούμε ότι είναι πολύ σημαντικές αυτές οι αποστολές, όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε όλο τον εκλογικό κύκλο και το έχουμε κάνει αυτό στην πράξη. Ξέρουμε ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση, όχι μόνο η στιγμή των εκλογών αλλά και το πριν και το μετά και θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε στο κείμενο. Τώρα, ε, ο Πατρίς ανέφερε Ε, ένα άλλο θέμα, ε, ο λόγος για τον οποίο έχουμε μειώσει τόσο πολύ τα ποσά είναι όχι για να καταστήσουμε πιο λιγότερο ευέλικτο το μέσο ε, γιατί ε, η υποστήριξη των τοπικών οικογένειων στη Βενγκάζι. ή ε, υγεία των γυναικών στη Λιβύη δεν είναι εμπιστευτικά πράγματα. Ε, αν μπορούμε λοιπόν να είμαστε ευέλικτοι σε ορισμένε περιπτώσεις, γιατί να μην ε, μοιραζόμαστε πληροφορίες με τους υπόλοιπους. Συνεπώς, θέλουμε ένα σχετικά υψηλό ποσό, αν ζητάμε ένα σχετικά υψηλό ποσό χωρίς ανάγκη να καταφύγουμε σε υποβολή προτάσεων και αιτήσει κλπ, αυτό θα πρέπει να το δικαιολογούμε κάθε φορά. Να είναι σαφές ότι χρειάζεται. Γιατί υπάρχουν ζητήματα δεν, στα οποία δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας, ακαιρεότητας κλπ. Ε, συμπληρωματική, όχι ιεραρχική αντιμετώπιση των δύο μέσων, πολύ σωστό. Ε, για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο έχουν δεσμευθεί έτσι ώστε να έχει προσθεμένη αξία, να συμπληρώσει κενά τα οποία αφήνει ο μηχανισμός ε, ανθρωπίνων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά θέματα, πρώτη ανάγνωση κλπ που θα μπουν τα των ε, πράξεων κατεξιοδότηση. Ε, θα το συζητήσουμε με τους σκιώδους και στο πλαίσιο των οριζόντιων ρυθμίσεων. Εγώ είμαι ανοιχτός. Αν θέλουμε να περάσουμε σε συμφωνία με στην πρώτη ανάγνωση, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε σίγουρα τη διαφάνεια. Τώρα, με χαρά μου άκουσα και δεν το ήξερα ότι υπάρχει πρόταση αύξησης του ποσού ε, του, από τα 100.000 στα 500.000 ευρώ ε, όταν χρηματοδοτούμε πολλά μικρο project δημιουργείται γραφειοκρατικό βάρος αν έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία ίσως μπορούμε τα project ε, ίσως μπορούμε να σημειώνουμε πιο γρήγορη πρόοδο. Ευχαριστώ πολύ για τις απόψεις σας, ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία σας τους ηγητές και τους αντιπροσώπους τους. Επίρα προτάσεις και από τους πράσινους, τις οποίες θα λάβω υπόψη. Αναμένω να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ Αλεξάνδερ και με αυτό ολοκληρώνεται αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Κατάθεση τροπολογιών, προθεσμία 14 Ιουνίου, 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας. Επόμενη ημερήσια διάταξη, οι ψηφοφορίες. Να περιμένουμε λίγα λεπτά. Να έρθουν οι συνάδελφοι. Έχουν ανακοινηθεί ε, για τις 12 ε, παρατέταρτο ε, οι ψηφοφορίες, οπότε διάλειμμα λίγων λεπτών. Λοιπόν, συνάδελφοι. Συνάδελφοι. Επόμενο θέμα στη μέση διάταξη είναι ψηφοφορία. Πολύ ιδιαίτερη ημέρα για μένα. Πρώτη φορά κάνω ψηφοφορίε. Παρακαλώ την επικοινωνία σα. <laughs> Uh, Θα ήθελα επίση να συγχαρώ τον κύριο Σαραφράγκα, δηλαδή να του ευχηθώ χρόνια πολλά γιατί έχει τα γενέθλιά του. Let's start uh, with the vote. Uh, we are going to... Ψηφίζουμε. Έκθεση για σύσταση στο Συμβούλιο για την 67η Γενική Συνέλευση, μάλλον σύνοδο της Γενικής συνέλευση του ΙΕ. Η τροπολογία 21 ψήφι Κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. Τώρα χρειάζεται έλεγχος, πιστεύω. Electronic check. Η ηλεκτρονική απολύθευση. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η συμβαστική παριθμόν 1 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εδώ χρειάζεται και πάλι έλεγχος. Παρακαλώ, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 29. It's closed. the vote. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η 30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 και 35 μαζί είπε Ναι, ταυτόσιμες. Κατά. Αποχές εγκρίνεται το σύνολο. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 2 σε 2 τμήματα. Τα εξής 3 Τμήμα πρώτο, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Το τρίτο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 41 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Η ηλεκτρονική απορρίθευση. Απορρίπτεται. Η 43 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Η 44 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται η 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ή 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές απορρίψετε 54 υπέρ κατά αποχές απορρίψετε 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 όχι διορθώνει ο πρόεδρος 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται χωριστή ψηφοφορία στην 66 τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα πάντα στην 66 υπέρ κατά αποχές δεν καταλαβαίνω. Έλεγχος για το δεύτερο τμήμα στην τροπολογία 66 βρετά. Πέρας. Απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ερχόμαστε στην 73 υπέρ. Α, όχι, έχουμε τη συμβιβαστική 4. Βιάστηκα, λέει ο πρόεδρος. Συμβιβαστική υπαριθμών 4. Your EPP. There's a problem with the EPP list. Yeah, in, in the EPP. I have the EPP list, yes. Α, κατάλογο του ΕΛΚ έχω εγώ. Και δεν γράφει εδώ συμβιβαστική 4. Ωραία. Πρέπει να ψηφίσουμε τη συμβαστική 4. Υπέρ. Against. Abstentions is... Ε, κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην 73. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 75. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 78 όχι. Ναι, 78 υπέρ, κατά αποχές δεν είναι σαφές ψηφίζουμε την 78 ηλεκτρονικά παρακαλώ πέρας εγκρίθηκε με μία ψήφο διαφορά 79 επέ κατά αποχές εγκρίνεται Η 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 5 υπέρ, συμβαστική, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 81, όχι. Πάμε στη συμβαστική 6 αμέσω υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 90 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 91 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος καλά. Για την 91 παρακαλώ. Απορρίπτεται με δύο ψήφους διαφορά. 93. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Νομίζω έχει απορριφθεί. 94. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 95. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 96. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και ερχόμαστε τώρα στην τροπολογία 97 σε τρία τμήματα παρακαλώ τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές και χρειάζεται ηλεκτρονική επαλήθευση ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα τώρα της τροπολογίας 97 Ακόμα τέσσερις συνάδελφοι πρέπει να ψηφίσουν. Πέρας. Εγκρίνεται. Με μία ψήφο διαφορά. Το τρίτο τμήμα τώρα της 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο για το τρίτο τμήμα. Η ηλεκτρονική απολύθευση. Τροπολογία 97 τμήμα τρίτο. Πέρας. Εγκρίνεται. 22-19 με 3 ψήφους διαφορά. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. No, no, 98. Για 98 μιλούσαμε. Την 98. 100. 100. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. 103 υπέρ, κατά, απόχέ. απορρίπτεται. 104 υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. 105 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 106 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται 107. Ποιος Λάινε. Αυτή η τροπολογία έχει αποσυρθεί. Νομίζω ότι ενημερωθήκατε. Όπως 35 και 36. Εγώ ήμουν ο ε, συγγραφέας αυτής και ε, συμφωνήσαμε να αποσυρθεί. 107. 135 και 136 έχουν αποσυρθεί. Θέλετε να πείτε ότι και οι υπόλοιποι συνυπογράφοντες έχουν ε, αποσύρει την ε, τροπολογία αυτή. Δεν είχα λάβει αυτή την, ε, αυτή την πληροφορία. Οι Άλβαρο, Μπρόκ, Κρέτ και λοιπά έχουν αποσύρει την υπογραφή τους. ο Λάμστορφ, γνωρίζω ότι τουλάχιστον ο κύριος Νταφ και ο κύριος Άλβαρο έχουν διατηρήσει τι υπογραφέ τους. Μακάρι να είχαν, να την είχαν αποσύρει. Δεν νομίζω ότι έχουν αποσυρθεί αυτές τι τροπολογίε. Δυστυχώ, θα πρότεινα και εγώ να έχει αποσυρθεί. Οπότε θα πρέπει να ψηφίσουμε την 107. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, συμβαστική 8 ε, σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίφθηκε, αλλά σε επαληθεύσουμε. And you're in favor against? Plus. Let's close the vote. Λήξη. Απορρίπτεται. Τμήμα 2 τη συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Επαλήθευση. Let's close the vote. Λήξη. Εγκρίνεται. Το τρίτο τμήμα εγκρίθηκε. Περνάμε στην 109. Πρέντα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 113. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 115 υπέρ συνάλφοι από το ΕΛΚ θα πρέπει να ψηφίσουν και αυτοί 115 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ηλεκτρονική ψηφοφορία so Uh 22 to 20 ε, εγκρίνεται γιατί ένα άτομο ψηφίζει χωρίς κάρτα 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 ηλεκτρονική επαλήθευση So please close the vote. Λήξη. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική παριθμόν 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφέ. Επαλήθευση, ηλεκτρονική επαλήθευση. Please close the vote. One more in Λήξη. Απορρίπτεται. 23, 23 κατά, 22 υπέρ. Οπότε, αφού απορρίφθηκε, Περνάμε στην 122 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές ηλεκτρονική επαλήθευση. Part, please. The vote is open. The vote is closed. Λήξη. Απορρίπτεται. 126. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 127. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 128. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 123. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται όχι απορρίπτεται 135 υπέρ 135 δεν την ψηφίσαμε την 135 κατά αποχές απορρίπτεται 136 Όχι, καταπίπτει. Απορρίφθηκε 135, άρα 136 καταπίπτει. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 11 λέει ξανά ο, ο πρόεδρος. 13. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14. Καταπίπτει 14. Όχι. Πρέπει να την ψηφίσουμε. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ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 κατά αποχές εγκρίνεται DVC υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Α, ηλεκτρονική επαλήθευση για το ΣΥ της ε, γνωμοδότησης της ε, Επιτροπής ΔΕΒΕ. Άλλοι δύο συνάλφοι. Ωραία. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. ΔΕΒΕ Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεβε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεβε όχι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται I υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Επαλήθευση, ηλεκτρονική επαλήθευση, δεν ήταν σαφές. Τρία ακόμη συνάλφοι δεν έχουν ψηφίσει. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Δεβε ΤΖΕΙ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεβε καίει Υπέρ. Κατά. εποχές, Εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο της έκθεσης. Please close. Δύο ακόμη συνάλφοι. Ίσως να φύγαν. Ε, εγκρίνεται με ευρία πλειοψηφία 39 υπέρ δύο αποχές. Καμία ψήφος κατά. Συγχαρητήρια στον κύριο Λάμστοφ. Έχουμε άλλη μία ψηφοφορία. Το ψήφισμα για τις διαπραγματεύσεις ε, για την ε, Συμφωνία Όπλων των Ηνωμένων Εθνών. Η συγκήτρια κυρία Τερμάκη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Τροπολογία 21 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 20 αποσύρθηκε, 19 υπέρ, κατά, αποχές, εκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 1 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές οι σοσιαλιστές δεν ψήφισαν η ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν για την 27 πέραση της ψηφοφορίας απορρίπτεται 28 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. 34. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ, κατά, άποχες εγκρίνεται, 38 υπέρ, κατά, άποχες δεν είναι σαφές, να κάνουμε μια επαλήθευση για το 38. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές απο, εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές επαλήθευση ε, παρακαλώ για την 50 Please close the vote. Πέραση ψηφοφορίας απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51 υπέρ. Όχι. Η 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απορρίπτεται αλλά για να το επιβεβαιώσουμε να κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα της 58. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 66 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα της 66 υπέρ, κατά, αποχές, ε, επαλήθευση. Πέραση ψηφοφορία, Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα του 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 67 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να κάνουμε έναν έλεγχο για την 68. Please close the vote. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές <laughs> απορρίπτεται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές να κάνουμε μια ηλεκτρονική παλήθευση για την 9.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 Πέραση ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 33 ψήφοι υπέρ, 2 αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Μία ανακοίνωση. Η επόμενη συνεδρία της Επιτροπής μας θα γίνει στις 4 Ιουνίου στις 5.30 το απόγευμα στις Βρυξέλλες. Καλή όρεξη. Okay.